Meine και κύριοι, να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μα και περνάμε πάρα αυτά στο σημείο 23 τη ε, ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για μια ε, ακρόαση για την έκθεση την οποία προετοίμασε η κυρία Φωτίγκα για τη στρατηγική επικοινωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τη προπαγάνδα εναντίον τη από τρίτου. Νομίζω ότι έρχεται στη σωστή χρονική στιγμή ε, το, η έκθεση αυτή. Γιατί σκόπα τη προπαγάνδα είναι να κατακτήσει τον εχθρό ε, χωρίς μάχη. Σε ό,τι αφορά την ε, προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, την ε, ριζοσπαστικοποίηση όχι μόνο εκεί αλλά και στις χώρες μας. Για να κερδίσουμε τη μάχη και τον πόλεμο θα πρέπει να κατανοήσουμε τις τακτικές ε, του αντιπάλου. Και θέλουμε να κατανοήσετε όλη τη σημασία αυτό. Γιατί θεωρώ ότι δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις και ξέρουμε ότι από τον πόλεμο του Βιετνάμ κανείς δεν έχει κερδίσει ε, πόλεμο χωρίς να έχει κερδίσει πρώτα τον πόλεμο της προπαγάνδας. Και είναι ο πόλεμος της εικόνας. Ε, γιατί δύσκολα μπορεί κανείς να καταπολεμήσει μια εικόνα, μια φωτογραφία. Εμείς ως δημοκρατικές ε, χώρες βρισκόμαστε σε μηνυκτική θέση σε σχέση με αυτοκρατικές χώρες, δικτατορικές χώρες που επικρατεί μία μόνο άποψη και η οποία και προβάλλεται στους λαούς αυτούς και στους άλλους λαούς. Γιατί προβάλλουν μια ιστορία επιτυχία την οποία εμείς δεν μπορούμε να προβάλλουμε γιατί έχουμε ε, μια ελεύθερη κοινωνία και δεν επικρατεί μια ε, άποψη αλλά πολλές. Και αυτό ο τελική ανάλυση είναι το πλεονέκτημά μας αλλά θα πρέπει να δεχτούμε να ιτηθούμε στον πόλεμο της προπαγάνδας και έτσι στον πλουραλισμό που επικρατεί στην κοινωνία μας θα πρέπει σήμερα να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα αυτή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, όχι μόνο προκειμένου να το πετύχουμε αυτό στις ε, περιφέρειες και στις περιοχές των άλλων, αλλά και στις δικές μας περιοχές, ε, για να κερδίσουμε τις ε, καρδιές και το μυαλό των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τη γίνεται στη Ρωσία σήμερα, βλέποντας με τα κοινωνικά μέσα, τα μέσα ενημέρωση, τα κανάλια και ναι. το... Η ΔΑΕΣ μέσω του διαδικτύου καταφέρνει να σταυτολογήσει κόσμο ε, στο Βέλγιο, στην Γαλλία, σε άλλες χώρες για να πολεμήσουν πόλεμο στη Συρία. Νομίζω ότι πολλοί δεν το έχουμε κατανοήσει ακόμα, αλλά βρισκόμαστε σε μία εποχή όχι ενημέρωσης, αλλά στρατολόγηση, στρατηγική επικοινωνία λοιπόν έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που κερδίζει κανείς και οι αντίπαλοι μας το κατανοούν αυτό και θα πρέπει να υπάρχει μία ε, ενιαία, ενωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα και να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε και σε ό,τι αφορά τις εκστρατείες προπαγάνδας από τρίτα μέρη. Γι' αυτό προσβλέπουμε λοιπόν σε αυτά που έχουν να μας πούν οι εμπειρογνώμονές μας που είναι ε, ειδικοί σε θέματα, ζητήματα. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Άντριου Ρέτσμαν, ειδικό ε, σε θέματα ασφάλειας ε, και εργάζεται και στο Πανεπιστήμιο της και γράφει και στο Guardian και σε πολλά άλλα μέσα. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τις ε, προοπτικές που έχουν να μας παρουσιάσει. Έχουμε τον κύριο Τζέρζι Μπομιάνσκι, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τη ρωσική προπαγάνδα στο σοβιτικό χώρο και θα ήθελα να μας μιλήσετε λοιπόν για τα απορίσματα του έργου αυτού και της σχετικής μελέτης που θα έχει αντίκτυπο και στις ε, ε, αποφάσει τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Και αυτό μεταξύ άλλων το έχει ζητήσει η κυρία Μογκερίνη. Και κατά τρίτον, τρίτο ε, παροσκεκλημένο και εμπειρογνώμονα, ο οποίο βρίσκεται μαζί μα μέσω τηλεδιάσκεψη, μια και δεν μπόρεσε να μεταβεί από τον Καναδά εδώ, ο κύριο Μομπίν Σάικ, ο οποίο είναι ειδικό σε θέματα ριζοσπαστικοποίηση και θέματα καταπολέμησης ε, της τρομοκρατίας και θέματα ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ας μας δώσουν λοιπόν τις πληροφορίες ε, που έχουν για την προετοιμασία της ε, έκθεσης της κυρίας Φωτίγκα. Πριν δώσω το λόγο στους ε, τρεις προσκεκλημένους, να ρωτήσω την κυρία Φωτίγκα αν θα ήθελε να πάρει το λόγο για να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Έχετε το λόγο κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και θα ήθελα εισαγωγικά να ευχαριστήσω και εσάς και τη Γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας για την διοργάνωση της ακρόασης αυτής και νομίζω ότι και οι τρεις ε, παρουσιάσεις έχουν εξαιρετική αξία για την προετοιμασία της έκθεσης. που θα παρουσιαστεί σύντομα για μια πρώτη εξέταση. Αντίθετα με τις προσδοκίες μας, οι γειτονικέ χώρες είναι εξαιρετικά δύσκολες και προς Ανατολάς και προς τον Νότο. Αντιμετωπίζουμε και τις όλο και πιο εχθρικές πολιτικές της ε, Ρωσίας πολύ εξειδικευμένε και επιτιδευμένες πληροφορίε για την ε, καταπολέμηση των θεσμικών μας, των θεσμών μας, των αξιών μας. Καθώς και πολύ επιθετική ριζοσπαστικοποίηση και σχετικές ε, στρατηγικές επικοινωνίας. Όλο και πιο δύσκολο να οριστούν, να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Στην έκθεση δε, την οποία και προετοιμάζω, θα αναφερθώ και στις δύο αυτές κατευθύνσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, αλλά σε ό,τι αφορά τη Ρωσία όλος ιδιαίτερος, μπορούμε να λάβουμε υπόψη και τη χρήση των πληροφοριών ως όπλο, γιατί επί μακρά χρονική περίοδο η χώρα αυτή χρησιμοποιεί τις ε, στρατηγικές επικοινωνίες ε, μαζί με τέτοιες ε, αμυγός στρατιωτικές τακτικές. Το παράδειγμα της Γεωργίας έχουμε, της Ουκρανίας, φυσικά όλος ιδιαίτερος, το οποίο αντιλαμβανόμαστε πλέον πλήρως ότι πριν την επίθεση στην Ουκρανία Και πριν δηλαδή την ε, επίθεση υπήρχε μια τέτοια στρατηγική. Σε ό,τι αφορά την ΝΤΑΕΣ τώρα, το Ισλαμικό κράτος, έχουμε ουσιαστική παρέμβαση σε ευρωπαϊκή επικράτεια από ριζοσπαστικοποιημένους νέους από όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά και κάτι λιγότερο, κάτι άλλο λιγότερο η καταπολέμηση των ε, δράσεών μας για τη διατήρηση της ειρήνης σε περιοχές ε, συγκρούσεων. Η στρατηγική επικοινωνία η οποία στρέφεται κατά των ειρηνευτικών μας αποστολών που σκοπό έχουν να διατηρήσουν μια κατάσταση ηρεμία και ειρήνη σε προβληματικέ περιοχέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω στι ε, παρουσιάσει που θα κάνετε. Ε, σα ευχαριστώ και το λόγο έχετε εσεί, κύριε Ρετμάν. γεια σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μπρόκ, που με καλέσατε. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για την προπαγάνδα πλευρά δημοσιογράφου ξεκινήσω με κάποιε παρατηρήσει για τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων εκδοχών των μέσων ενημέρωσης και την, των ε, παρακινήσεων για λόγους μίσους κλπ. Και, και μετά θα δούμε και το Ολλανδικό δημοψήφισμα για την Ουκρανία και δείξουμε πόσο μπορούν οι απόψεις των μέσων ενημέρωσης να επηρεάσουν αρνητικά τις εξελίξεις και να εκφράσω ιδέες για τις ευρωπαϊκές αρχές και τι μπορούν να κάνουν τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για αντίδραση. Καθοδόν θα εκφράσω και κάποιες σκέψεις για άλλες μορφές προπαγάνδας ή διαμόρφωση των ειδήσεων από τα εύσιλον, κυρίω από την νότια γειτονιά τη Ευρώπη και πώ χρησιμοποιεί το Ισραήλ τα ΜΜΕ για να προωθεί του στόχου του όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Τι εννοούμε αυτό άποψη που εκφράζουν τα μέσα. Ο ορισμό τη λέξη πριν που χρησιμοποιώ για αυτό το που θα προσπαθώ να πω είναι ότι προωθούνται μέσω προπαγάνδας μηνύματα ούτω ώστε να δημιουργήσουν διανοητική και συναισθηματική αντίδραση που εξυπηρετεί κάποια ομάδα συμφερόντων. Άρα αυτό διαφοροποιείται από την κανονική κάλυψη γεγονότων που ενημερώνει το κοινό για να αποφασίσει το κοινό το ίδιο. Δεν υπάρχει κάτι που είναι 100% αντικειμενικό στη δημοσιογραφία. Ε, Κάποιο ε, που γράφει ένα άρθρο έχει κάποιε υποθέσει μέσα του. Μιλάω όμω για συνειδητή συστηματική εκστρατεία με συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Όλοι γνωρίζουν όταν το βλέπουν αυτό ότι είναι κάτι τέτοιο, ότι είναι μια προπαγάνδα. Μπορείτε να το καλέσετε προπαγάνδα. Εγώ το ονομάζω άποψη δια, ε, διαμόρφωση τη εικόνα, spin στα αγγλικά. Το βλέπετε και, σε κάποια, και στα ρωσικά ΜΜΕ και στα δεξιά Ισραηλινά μέσα. Το Daily Mail, το Daily Express παρουσιάζουν οποιασδήποτε ειδήσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με τέτοιο τρόπο για να ξεκινήσουν ε, να κερδίσουν ψήφου για την εκστρατεία για να αποχωρήσει ε, η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή τα μέσα τα αντίστοιχα τεσδινά κινούνται κατά τη Παλαιστίνη και τα ρωσικά ΜΜΕ δείχνουν με κακό φως το, τη Δύση. Ε, η υπηρεσία Sputnik ε, προσπάθησε να παρουσιάσει τη δική τους άποψη για την κρυμμένη στην Ευρώπη. Μου έστειλε δωρεάν υλικό και εικόνες και 30% των πολιτών θεωρεί αυτή ε, η υπηρεσία ότι θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι ανοίξει η Ρωσία. Τώρα εξαρτάται πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Όπως ε, και τον πόλεμο στη ροή της Γάζας. Ε, έλεγαν ότι σκοτώθηκαν εκατοντάδες Παλαιστίνοι και λίγοι Ισραηλινοί κάποια μέσα ενημέρωσης. Η ρωσική άποψη είναι διαφορετική. Ελέγχεται, χρηματοδοτείται το Κρεμλίνο. Και υπάρχουν διάφορες ειδήσει που διαδίδονται στο διαδίκτυο. Η κλίμακα και η φύση του προγραμματισμού του ρωσικού είναι μοναδικό στο είδος του. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά όμως με τον τρόπο που κινούνται τα ΜΜΕ. Λοιπόν, επεκρινόταν η κυβέρνηση Κατσίνσκι στην Πολωνία και άλλες κυβερνήσεις αλλού. Και βλέπαμε επιθέσεις στα κοινωνικά μέσα. Σαν να ήταν οργανωμένη όλη η επίθεση και η διάδοση στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα. Θέλουν να δημιουργήσουν αισθητική αβεβαιότητα οι Να δείξουν ότι τι κυβερνήσει και όλα τα ΜΜΕ ψεύδονται, οπότε δεν υπάρχει κάποια αντικειμενική άποψη για να ενημερωθεί κανεί. Η ρωσική Πρασβεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμαρτύρεται και μου λέει ότι λέω ότι υπάρχουν στρατεύματα ρωσικά στην Ουκρανία χωρί να λέω ότι είναι η δική του θέση ότι δεν υπάρχουν στρατεύματα ρωσικά. Θέλουν να, να αντιστρέψω τα γεγονότα προς χάρη του πλουραλισμού. Ε, μία ΜΚΟ στο Ισραήλ με έφερε στην Ιερουσαλήμ δείχνοντας ότι δεν παραβιάζει το Ισραήλ το διεθνές δίκαιο διότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Αυτή την άποψη να προωθήσουν όταν ε, τελικά όταν έπεσε το αεροπλάνο η πτήση MH17 και λέγαμε ότι έφταιγε η Ρωσία, αυτοί θα αναπαρουσίσουν δική του έρευνα. Επίση, όταν γίνονται κάποιε βιοπλαγίε από πλευρά Ισραηλινών στρατιωτών, οι Ισραηλινοί θέλουν να ανθώσουν του στρατιώτε. Η Daily Mail ε, παρουσιάζει το ευρωσκεπτικιστικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να είναι βραβερό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι Ρώσοι θέλουν να νομιμοποιήσουν μια τρομακτική δικτατορία που άρπαξε την Ουκρανία και έχει προξενήσει τουλάχιστον 1.000 θανάτου. Δεν είναι όμως παρακίνηση κλιματικής φύσης αυτή. Το Σύνταγμα τον είπα προστατεύει την ελεύθερη έκφραση, όπως και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλά είναι έγκλημα στη ΣΥΠΑ να παρακινήσεις βιοπραγία αν αυτό γίνει ε, παρουσιάζοντας μια αξιόπιστη απειλή ότι μπορεί να γίνει. Η προπαγάνδα του Ντάις οδηγεί σε διαφόρους να πάνε ε, στη Συρία ε, και τους πείθει για τον σκοπό. Δεν δημοσιεύεται email ψευδεί ειδήσει σε τέτοιο βαθμό, παρόλο που έχει μια κλίση. Και τα ζενά μέσα προσπαθήσουν να δώσουν μια πάνθρωπη εικόνα των Παλαιστινίων, αλλά κανείς δεν συγκρίνεται με την παρακίνηση των Ρώσων να στραφούν κατά των Ουκρανών. Δεν υπάρχει ε, κα χρόνος να παρουσιάσω όλα τα ψεύδη. Λοιπόν, η ρωσική προπαγάνδα για τη μεταστατική κρίση πλησιάζει αυτή την εικόνα παρουσιάζει την προπαγάνδα όπως η κοπέλα που βιάστηκε στη Γερμανία. Και ε, επίσης τις διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στη Γερμανία, που μπορεί να οδηγήσει αυτή η παρουσίαση της, του βιασμού κλπ. να κινηθούν οι άνθρωποι στη Γερμανία κατά των μεταναστών. Συνάδελφός μου Ολλανδός κάλυψε τα γεγονότα στο Άμστερνταμ. Μίλησε με πολλούς στον δρόμο και στους σταθμούς που επανέλαβαν ότι Έλεγαν οι Ολλανδοί ότι η Ουκρανία ανήκει στη ε, επιρροή τη Ρωσία, είτε μα αρέσει είτε όχι. Άλλοι είπαν ότι διεφθαρμένη χώρα η Ουκρανία. Αλλά οι συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Αυτό δεν το είπαν. Στι γεωπολιτικέ συζητήσει για σφαίρε επιρροή δεν υπάρχει αλήθεια. Η Ουκρανία μπορεί να είναι διεφθαρμένη. Όμω, οι Ρώσοι κυκλοφορούν και ψευδείς, ψευδή βίντεο Ουκρανών φασιστών που απειλούν να ανατινάξουν τους Ολλανδούς αν ε, όχι στο δημοψήφισμα. Τι να κάνουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δύο πράγματα. Η δηλαδή αυτή η κυψελίδα, ε, η κυψέλη καταπολεμήσεως της προπαγάνδας. Ή το ED, ούτως ώστε να παρουσιάσουν αντίθετο αφήγημα που θα εκπέμπουν. Ελάχιστα αυτά χρήματα που δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια των εκατομμυρίων που δαπανούν οι Ρώσοι. Βοηθά όμως η προσπάθεια. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να εξετάζουν το Stratcom ή να βλέπουμε ποια ψεύδι λένε οι Ρώσοι. Για το ED τώρα. Το κυβερνητικό υλικό τελικά δεν είναι μερόληπτο. Ο κύριος Παμανόφσκι, αυτό πώς θα το αντιμετωπίσει. Έχουμε τρεις αντιδράσεις. Πρώτα όσον αφορά την παρουσία των γεγονότων με μια απόχρωση. Πολιτική αντίδραση και να στηρίξουμε και τα φυστάμενα μέσα ενημέρωσης. Για τα πατηλά στοιχεία, ρυθμιστική επίθεση θα έλεγα εγώ, κατά των παρανόμων αυτών ειδήσεων. Στο πρώτο στοιχείο δεν πρέπει να επαναφεύρουμε τον τροχό. Έχουμε καλέ δομέ. Μπορούν να αντιδράσουν στα εχθρικά μηνύματα χωρί να επηρεάζεται την κοινωνικότητά μα. Τα βασικά πολιτικά κόμματα έχουν προγράμματα, αξίε. Ίσως δεν ήταν κατά ενεργά τα κόμματα να προβάλλουν το αντίθετο μήνυμα αυτών των Ρώσων. Το CDU στη Γερμανία, οι σοσιαλιστέ στη Γαλλία, οι συντηρητικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν. Προσπαθούν να επανεκλεγούν και εξοδεύουν ενέργεια και χρήματα. Αν έκαναν προσπάθειε να εξηγήσουν τι γίνεται στην Ουκρανία και τι γίνεται στη Ρωσία, αν κάναν την ίδια προσπάθεια όπω κάνουν να επανεκλεγούν, θα κινούνται προ την κατεύθυνση τη σωστή. Και στην Ολλανδία δεν υπήρξε σωστή υποστήριξη για το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Είπαν στη Γερμανία ότι και αντίθετοι ε, προς το όχι, δεν κινήθηκαν αρκετά στην Ολλανδία. Για λόγους ε, ψηφοθυρικούς. Και κάποιοι για τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις ε, πηγαίνουν και ζητάνε χάρες από τη Ρωσία ή καλομεταχειρίζονται τη Ρωσία για λόγους οικονομικούς. Ο Λάντκι Μέρκελ Φερρυπίν ε, όταν επετέθηκε η Ρωσία στην Ουκρανία δεν κατονόμασε τη ρωσια για λογους οικονομικους ο λαντκι μερκελ φερρυπιν οταν επετεθηκε η ρωσια στην ουκρανια δεν κατονομασε τη ρωσια σαν την επιθετική δύναμη. Η του Today, το κανάλι αυτό, παίρνει πολλά χρήματα από τη Ρωσία. Αλλά υπάρχουν χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική που μπορούν να αντιδράσουν, διαθέτοντα όμω κατάλληλου πόρου. Θα πω αυτό που είπα και προηγουμένω σε άλλε φάσει. Έχετε ευθύνε, διαμορφώνετε τι γνώμε. Αποφασίζοντα λοιπόν για την αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωση στην Ουκρανία οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στη, στην έκδοση των κειμένων των εφημερίδων. Το Ταν Γιούγκ, πάρω παράδειγμα. Η υπηρεσία, το, το πρακτορείο ειδήσεων της Ιγκοσλαβίας χρεοκόπησε διότι δεν βρέθηκε αγοραστής. Ταυτόχρονα η υπηρεσία Σπούτνικ της Ρωσίας ξεκίνησε εκπομπές στα σερβικά. Έχουν και στο διαδίκτυο. Στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα στη Μητρόβιτσα. Ε, εκεί γίνονται εκπομπές ρωσικής προπαγάνδας και παρακινούν σε εθνοτική βία. Και αρχές του Φεβρουαρίου με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, δολοφονούν τάχα εθνοτικούς Σέρβους στο Κωσυφοπέδιο. Και δεν πρέπει να υπερικόπτονται δηλαδή οι εκπομπές σε γλώσσες. Έχουμε ρυθμιστικές πιέσεις. Κινήθηκαν οι Βρετανοί κατά του του Today. Οι Γερμανοί ε, κινούνται κατά εκείνων που παρουσιάζουν την εικόνα της κοπέλας που βιάστηκε κλπ. Θα πρέπει να κινηθούμε κατά, της, ε, κατά του Δημήτρη Κασίλιεφ που διαδίδει προπαγάνδα. Χρειάζεται όμως καλύτερο συντονισμό και όχι μεμονωμένες κινήσεις. Έχουμε νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καιρότητα των μέσων ενημέρωση. Οι συνάδελφοι στο πάνε θα πούν περισσότερα. Όπω η οδηγία για τα οπτικοακουστικά. Γιατί να με επικαιροποιηθούν τα μέτρα. Να γίνει συντονισμένη προσπάθεια. Να εφαρμοστούν τα μέτρα. Πώ παγώνουμε εκείνου που παρακινούν τη ριζοσπαστικοποίηση στην Ισλαμιστική, αλλά αγνοούμε εκείνου που κάνουν παρόμοια παρακίνηση για δολοφονίε και δια, ε, βασανιστήρια στον Ντομπά. Γιατί τα Υπουργεία μα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει διαπιστευτήρια τύπου σε εκείνου που δεν έχουν καλό ιστορικό και εφευρίσκουν ιστορίες ε, προς εξυπηρέτηση του Κρεμλίνου. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Προσβλέπω στις ερωτήσεις σας. Now Ζέζι Πιομιανόφσκι τώρα λέει ο πρόεδρος. Με αυτό το όνομα νομίζω θα έχω προβλήματα σε όλη μου τη ζωή. Ζέζι έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Έλμαρ. Να, φαίνεται πως γίνονται επικαλύψεις ε, στη δουλειά μας. Μια που ε, σε αυτόν τον φορέα για τη δημοκρατία είναι ο Έλμαρ ε, πρόεδρος, οπότε βλέπουμε ότι σε αυτές μας προσπάθειες έχουμε πολλαπλές ιδιότητες. Και θεωρούμε, όσον αφορά το φορέα μας, ότι πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια δεν μπορώ παρά να συγχαρώ την ε, κυρία Φωτίγκα για το έργο της. Έχουμε τόσους Ευρωπαίους πολιτικούς που προσπαθούν προς την κατεύθυνση, οπότε αυτό σημαίνει το θέμα θα πρέπει να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα. Τώρα θα πρέπει να ε, πούμε αυτή την ε, γνωστή επιφύλαξη που αφορά την προπαγάνδα και αυτό νομίζω ότι αφορά την προπαγάνδα και πιστεύεις ότι η στρατηγική επικοινωνία είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Γιατί και εμείς το EED, ε, σε αυτόν τον φορέα για τη δημοκρατία στην Ευρώπη, βλέπουμε τα πράγματα από την οπτική γωνία των δημοκρατικών αξιών και των βασικών ελευθεριών. Και η επικοινωνία αλλά και ο αγώνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, Πολλέ φορέ ε, επικαλύπτονται, παρόλα αυτά όμω είναι δύο διαφορετικέ γωνίες. Ε, το EED, η οφορία μα δεν εμπλέκεται σε στρατηγική επικοινωνία καθεαυτή. Επίση, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα τοπικά μέσα ενημέρωση, να αποκτήσουν τι δυνατότητε που πρέπει ούτω ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν και να γίνουν ανεξάρτητα ποιοτικά ΜΜΕ και επίση να αποτελούν διάβλου επικοινωνία και ένα μηχανισμό προστασία δημοκρατικών αξιών. Οπότε σε σχέση με αυτό θα σας πω ότι ό,τι βοήθεια και να δοθεί δεν θα πρέπει να πειράξει την έκδοση του εντύπου ή να προτείνει ε, το πώς θα κάνει τη δουλειά της ε, αυτή η εφημερίδα, το ΜΜΕ ή οποιαδήποτε δημοσιογραφική δραστηριότητα και Άρα θα πρέπει η πληροφορία να γίνει όσο καλύτερα μπορεί το, το μέσο ενημέρωση. Επίσης κάτι το οποίο δεν έφερε και ο πρόεδρο μα Πέρσι ο φορέας μας έκανε ένα συντονισμό για να γίνει μια μελέτη βιωσιμότητα ε, ε, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο 2015 που αφορούσε τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό ήταν ε, παραγγελία της Ολλανδικής κυβέρνησης και ήμασταν κάτι σαν διαμεσολαβητή μεταξύ κυβερνήσεων και σχεδόν των πολιτών. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον φορέα μα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ήταν αυτό κάτι καινούργιο, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια υποστηρίζουμε ανεξάρτητα ΜΜΕ στι χώρε, της γυρνιάζουσε με την ε, Ευρώπη και είναι αυτό μία από τι βασικέ μα δραστηριότητε. Ξεκινούμε λοιπόν από Ανατολά και θα πρέπει εδώ να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά, να δούμε ε, την περιπλοκή που προκύπτει από την προπαγάνδα του ρίσκου κράτους και κατόπιν προχωρούμε προς νότον και θα διατυπώσουμε και κάποιες συστάσεις. Όσον αφορά την Ανατολή τώρα σήμερα, αυτό το οποίο ε, βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ολοκληρωτική κυριαρχία των φωνών που είναι στο μήκος κύματος του Κρεμλίνου. Αυτό δεν είναι καινούριο. Και ε, θεωρούν εκεί ότι ο πολιτικός έλεγχος είναι ένα μέσο εξωτερικής πολιτικής. Ο Πούτιν ακούσε μια δρομή 12 ετών για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και κάνουμε τώρα μια αναδρομή στο παρελθόν, όχι πολύ παλιά, έχουμε ε, την κατάληψη του πόρταλ της διαδικτυακής πύλης lenta.ru το 2014 και επίσης έπαψε να έχει ανεξαρτησία το πρακτορείο Ρία Νόβοστη το 2013. Οπότε υπήρχε ε, ε, θέση υπό διαχείριση και καθάριση των μέσων αυτών και βλέπουμε ότι η Ευρώπη και γενικότερα η Δύση κλείσαν τα μάτια. Και μετά είχαμε τον πόλεμο στην Κρυμαία στην στην Ουκρανία, είχαμε την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας, οπότε η Ευρώπη ε, τότε κατάλαβε ποια είναι τα αποτελέσματα της κρατικής προπαγάνδας. Ήταν αυτό ένα σημείο καμπή, αλλά επίσης με το και ένα καινούριο κεφάλαιο στην πολιτική πληροφορία της ε, Ρωσίας και από τότε έχουν ποικιλία μέσων και προσπαθούν επομένως να έχουν μια εργαλειοθήκη που ασχολείται και με το διαδίκτυο και μέσα γενικής δικτύωσης, δηλαδή τα, τα φόρουμ σαν πολλαπλασιαστικούς ε, παράγοντες, αλλά και το τρολάρισμα. Οπότε τώρα έχουμε ε, κάποια άλλα μέσα που θέλουμε να στηρίξουμε όσο αφορά την εξαρτησία τους και είναι ρωσόφωνα και βρίσκονται στις χώρες της Ανατολικής Τερικής Σχέσης. Και αυτή η έκθεσή μας, αυτή η μελέτη μας ε, είναι γνωστή σε εσά. Οπότε απλώ θα σταθώ σε κάποια επιχειρήματα μόνο. Γιατί επιβεβαιώθηκε με τη μελέτη αυτή ότι τα ρωσόφωνα μέσα αλλά και οι αναγνώστε στα ακροατήρια ε, είχαν εγκαταλειφθεί, είχαν παραμεληθεί, ε, ούτε υπήρξαν επενδύσεις και έτσι το Κρεμλίνο πάρα πολύ εύκολα έκανε τη δουλειά του. Οπότε αυτό ήταν το αποτέλεσμα των εξή. Πρώτον, προσβασιμότητα και κυριαρχία των πηγών που μεταδίδουν και διαβιβάζουν τα μηνύματα του Κρεμλίνου στους ρωσόφωνους αλλά και στους ξένους. Οπότε βλέπουμε το εδώ πέρα ε, το πιο βασικό μέσον είναι η τηλεόραση και δεύτερον έρχεται το ίντερνετ δια τηλεφώνου και έτσι κυριαρχούν στους ε, ακροατές ε, για τα νέα και για τη διασκέδαση. Και έτσι έχουμε το κανάλι Russia Today, το Russia Direct και το Russia Beyond the Headlines. Γιατί βλέπουμε όμως ότι αυτά τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι ο μόνος τρόπος να περάσουν οι ρωσικές απόψεις στη Δύση. Γιατί έχουμε επίσης και άλλους φορείς όπως ε, δημοσιογράφους που ε, πληρώνονται από το ρωσικό κράτος Έχουμε ομάδες προβληματισμού, think tanks, έχουμε λομπίστες κλπ. Και ε, βλέπουμε ότι πάρα πολλά χρήματα διατίθενται για αυτούς τους ε, σκοπούς. Αυτό είναι βέβαια καλό νέο. Ε, πάντως η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής πέρα από τους ρωσόφωνους είναι περιορισμένη. Τώρα αφορά την διασκέδαση είπαμε ότι υπάρχει κάποιο είδους ε, συναισθηματική ε, αφήγηση γιατί υπάρχει κάποιο είδου νοσταλγία για το, το παρελθόν, ιστορικά έργα. Ε, επίσης παριστάνουν τα θύματα ε, ο ρωσόφωνος πληθυσμός σύμφωνα με αυτά τα μέσα και οπότε επειδή είναι συναισθηματικά φορτισμένα ελκύουν την προσοχή και έχουν και ποιοτικέ παραγωγές πάντως. Και ξεκάθαρο προήψε ότι η προπαγάνδα και η αντιπροπαγάνδα τελικά ε, μείωσε την εμπιστοσύνη ε, προς τα ΜΜΕ. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν αποδίδει αποτελέσματα εκεί. Να δούμε τώρα δύο βασικά χαρακτηριστικά του γιατί είναι τόσο αποτελεσματικό αυτό το, το υλικό που κατασκευάζεται στο Κρεμλίνο έχουμε τον κύριο Πομεράντζικ ο οποίος μας βοήθησε σε αυτή τη μελέτη βασικά αυτό το οποίο θα εντοπίσουμε τώρα είναι την παραγωγή από το Κρεμλίνο ενός παράλληλου κόσμου με εξειδικευμένες ε, περίπλοκες ε, ε, κατασκευή, κατασκευή πληροφοριών, με παραπληροφόρηση, με χειραγώγηση, με ψέματα και τελικά ε, αυτό το οποίο περιγράφουν είναι ότι η Ρωσία είναι υπό ε, ε πολιορκία και ότι για να μπορέσει να επιβιώσει θα πρέπει κανείς να δείξει πίστη προς τον αρχηγό του φρουρίου, τη Ρωσία δηλαδή. Και βλέπουμε τι γίνεται με τις βασικές αξίες της δημοκρατικές, για το κράτος δικαίου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και εδώ και η διάσταση της ασφάλειας, αλλά υπάρχει και θέμα της στρατιωτικής ασφάλειας των ε, γειτόνων μας και η δική μας ασφάλεια. Οπότε είναι λάθος κανείς να θεωρείται αυτή η προπαγάνδα και αυτή η χειραγώγηση των μέσων είναι κάτι το απομονωμένο. Θα πρέπει αυτά να τα δούμε μέσα στο ευρύτερο σκηνικό. Είχαμε μια ανάλυση πρόσφατη του κέντρου Λεβάντα και είδαμε ότι συνέχεια όλο ένα και περισσότερο γίνεται αποδεκτή ως πιθανή λύση στα προβλήματα ο πόλεμος. Αυτό γίνεται στην ρωσική κοινωνία και εδώ μιλούμε για την καρδιά και το μυαλό εκατομμυρίων οι οποίοι ζουν στην ίδια ήπειρο με εμάς. Εάν αυτό δεν είναι μια σοβαρή απειλή, τι είναι τότε. Precisely the επειδή είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα, αυτό που χρειάζεται είναι μια αντίδραση ευφύης και καινοτόμα. Δηλαδή, εδώ εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά θα πρέπει ο καθένας να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί και να την αναλάβει. Τώρα, για το ίδιο το φορέα μας το βασικό μας ζήτημα ήταν τι γίνεται με το ακροατήριο το ρωσόφωνο και είπαμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τα ρωσόφωνα μέσα στην, στις χώρες ανατολικής τερικής σχέσης και έτσι να διορθώσουμε την ανισορροπία και το ότι παραμελήσαμε και ξεχάσαμε αυτά τα μέσα. Αλλιώς πρόκειται να χαθεί και άλλη γενιά ρωσόφωνων από την χειραγώγηση των ε, Ρώσων. Ε, οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να ανακτηθεί η μισθοσύνη προς ε, τα τοπικά ΜΜΕ και ε, θα πρέπει ο κόσμος να ελκυστεί προς αυτά αν αυτά τα μέσα θίγουν ζητήματα της καθημερινής τοπικής ζωής. Επίσης είπαμε ότι έχουμε διπλή προσέγγιση πρώτα-πρώτα να ενισχύσουμε τα ανεξάρτητα μίντια και ταυτόχρονα θα πρέπει να επενδύσουμε σε κάποιες πλατφόρμες συνεργασίας και θα πρέπει τελικά αυτά τα μέσα να έχουν κάποιο είδους μακρόπνοη υποστήριξη από τους διεθνείς δωρητές. Άρα πρόκειται για μια ε, προσπάθεια με συνεργασία. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς μια με αμοιβαία ε, ενίσχυση, με συμπληρωματικότητα και με συντονισμό των δωρητών θα μπορούμε να έχουμε οικονομίες κλίμακας και με αυτή την προσέγγιση να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ε, απόδοση αυτών των μέσων. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την ποιοτική δημοσιογραφία, πλουραλισμό και θα πρέπει να τους αφήσουμε, τους ρωσόφωνους, να προβάλλουν και να παραγάγουν ό,τι θέλουν. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τάσεις, να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες ε, αυτού του κοινού και να δούμε το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στις οικονομικές αποφάσεις ε, των ε, επενδυτών του ιδιωτικού τομέα. Βέβαια στη Ρωσία θα έχουν πάρα πολλές δυσκολίες να επενδύσουν και πάρα πολύ ανταγωνισμό, αλλά μπορεί να ενεργήσουν αυτοί οι επενδυτέ σε άλλε χώρε που έχουν ρωσόφωνο πληθυσμό. Αυτέ είναι οι συστάσει τη έκθεσή μα. Και τώρα για να στραφούμε προ Νότον, εκεί επίση ε, υπάρχει προπαγάνδα γιατί αυτό έγινε από το Ισλαμικό κράτος και ανταγωνίζεται περίεργως την ρωσική κρατική προπαγάνδα. Βέβαια είναι δύο χωριστά ζητήματα αυτά και έχουν λίγα κοινά σημεία γιατί υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές, έχουμε ένα κράτος όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από το κέντρο και από την άλλη μεριά έχουμε ε, το, το, το Ισλαμικό κράτος που δεν είναι κανονικό κράτος και έχει διάφορα κέντρα εξουσίας. διαφορετικές μεθοδολογίες ο καθένας, αλλά μοιάζουν. Η μεγαλύτερη όμως διαφορά των μεν από τους δε είναι στον αντίκτυπο, ιδίω μέσω και μακροπρόθεσμα. Η προπαγάνδα του Ισλαμικού κράτους έχει τακτικό χαρακτήρα, είναι κάτι το περαστικό και δεν αποτελεί συστημικό πρόβλημα η προπαγάνδα του ρωσικού κράτους είναι πολύ πιο επικίνδυνη γιατί αποτελεί ε, κάτι το στρατηγικό, κάτι το που έχει διαρθωτικό δομικό χαρακτήρα. Ανοίξουμε μια ματιά στην ρωσική προπαγάνδα θα δούμε ότι επηρέασε εκατομμύρια προσώπων και συνεχίζει να είναι θέμα συζήτησης. Τώρα, εάν έχουμε 5.000 μαχητές που τους ε, επιστρατεύει για να πολεμήσουν στη Συρία ε, το ιστορικό κράτος ή θέλει να τους στείλει εδώ να γίνουν τρομοκράτες, συζητούμε ότι αυτό είναι καταστροφή. Άρα θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους ε, διάσταση. Μην υποβαθμίζουμε το ένα έναντι του άλλου. Οπότε, από αυτής της πλευράς, για να δούμε ποιες είναι οι βασικές συστάσεις όπως λοιπόν οι ειδικοί. Πρώτα-πρώτα να στηρίξουμε τα ανεξάρτητα μίντια. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε. Εκεί θα πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο. Ξέρουμε ποιο είναι το κοινό αυτών των ε, μέσων ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται να τους καθοδηγήσουμε για την καθημερινή που θα ακολουθήσουν. Αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να μείνουν αυτά τα μέσα ανεξάρτητα. Βέβαια θα πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει συνειδητοποίηση στις κοινωνίες και βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται όσον αφορά τις δημοκρατικές αξίες και αυτό το ε, άρα εκπαίδευση και συνειδητοποίηση των κοινωνιών. Ε, επίσης θα πρέπει να ξεμπροστιάσουμε ε, την παραπληροφόρηση της Ρωσίας σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες που ε, διαδίδουν ψέματα στις δικές μας χώρες και στη δική μας χώρα. Εδώ έχουμε πολλά μέσα νομικά, ηθικά και έχουμε και επίσης μεθόδους ανείγνευσης παρανόμων χρημάτων, τέλος των βρώμικων χρημάτων, προϊόντων εγκλήματος που υποστηρίζουν αυτά τα παραπλανητικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος, κύριε Πομιανόφη, σας ευχαριστούμε. Και τώρα τον λόγο θα έχει ο κύριος Σάικ, ο οποίος είναι ειδικό για την απορριζοσπαστικοποίηση και στα θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας και στα θέματα της ε, ασφάλειας. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Έχει συγγράψει μια σειρά βιβλίων. Πριν από 20 χρόνια περίπου είχε πάει σε Ινδία και Πακιστάν και είδε πώς γίνεται εκεί η στρατολόγηση και κατόπιν είχαμε τις τρομοκρατικές ενέργειες ε, της 11 η Σεπτεμβρίου. Τότε αναθεώρησε τις απόψεις του. Πήγε στην Συρία, μελέτησε από κοντά ε, τον ε, Ισλαμισμό, απορριζοσπαστικοποιήθηκε το 2004, πήγε στον Καναδά, οπότε και εξειδικεύθηκε στα θέματα τα οποία My, my and blessing to, to be addressing uh, the parliament in Brussels. Σας ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή που ε, έχω την ευκαιρία να μιλήσω προς το Κοινοβούλιο στην Ευρώπη. Να σας πω ότι εργάστηκα δύο χρόνια undercover ε, και σε πολλές περιπτώσεις ε, έκανα ε, και online και στην πραγματική ζωή και ε, κατέθεσα σε δικαστήριο. 2010 όταν ε, ολοκληρώθηκαν οι δικαστικές υποθέσεις μπήκα στο Twitter και στο Facebook και είδα ότι πολλοί νέοι συζητούσαν τα θέματα αυτά που είχαν να κάνουν με τη θρησκεία, που είχαν να κάνουν με τα παγκόσμια περιστατικά. Είχε ξεκινήσει το 2010 ο πόλεμο στη Συρία, Αραβική Άνοιξη 2011-2012 και οι συζητήσει των νέων να πάνε στην Συρία να πολεμήσουν ε, άρχισαν να γίνονται όλο και πιο συχνές και είδα να ανθεί ε, στο διαδίκτυο η νεολαία αυτή του ίσης το 2012, 2013, 2014 και το 2015 σε μεγάλο βαθμό. Σχεδόν καθημερινά ήμουνα σε επαφή με αυτή την νεολαία του ίσης και είχα διάφορες προσεγγίσεις που θεωρούσα ότι ήταν ωφέλιμες και που θεωρούσα ότι αν τις είχα εφαρμόσει στους νέους θα ήξερα τι δουλεύει και τι όχι. Τότε λοιπόν άρχισα να ακούω σε διάφορες διασκέψεις ε, θέματα ριζοσπαστικοποίησης πολλού συμπεριογνώμονες ε, που είχαν πέσει από τον ουρανό, από ό,τι φαίνονταν τέτοια εντύπωση έδιναν και μιλούσαν για τη ριζοσπαστικοποίηση. Τους παρακολούθησα λοιπόν για να δω κατά πόσον ήταν αποτελεσματική σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που περνούσαν προς τους νέους αυτούς. Καταρχάς, λοιπόν, η προσέγγιση μου ήταν η εξή. να χρησιμοποιώ τις Ισλαμικές πηγές για να καταπολεμήσω την προπαγάνδα της ΔΑΕΣ. Και κάτι στο οποίο είναι πολύ καλή η ΔΑΕΣ είναι να διαλέγει από το Κοράνι κάποια αποσπάσματα και τα οποία και χρησιμοποιούν για τους σκοπούς τους, τα οποία δίνουν και ένα πακέτο, τα οποία θα συνοδεύουν και με ένα πακέτο πάρα πολύ ε, εξειδικευμένο σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωση και έτσι για τους νέους ο συνδυασμός αυτό μαζί με κάποια τραγούδια ε, έχει μεγάλο αποτέλεσμα και αντικτύπο. Τρομοκρατία λοιπόν με ισλαμικό κουστούμι, με ισλαμική ε, μεταμφίεση. Τρομοκρατία με ισλαμική μεταμφίεση. Έτσι θα το περιγράφα. Και κάτι που ανακάλυψα ήταν ότι δούλευε και η τους, είχε αποτελέσματα και μπόρεσα να έρθω σε επαφή με μέρη της, ε, του Ίσης, ακόμα και με τη Αλκάιντα. Μπορούσα να τους μιλήσω σε μια γλώσσα που καταλάβαιναν και να χρησιμοποιήσω το ίδιο Κοράνι και να ε, έχουμε επιχειρήματα και αντιπιχειρήματα και μια έτσι τέτοια επικοινωνία. Όταν σας λέω ότι πρόκειται για ένα βαρέλι με ιδέες, όταν το λέμε αυτό, θα πρέπει να το εννοούμε. Θα πρέπει να είμαστε και να επιμένουμε στις αξίες μας, να είμαστε σταθεροί και να προκαλούμε τα δικά τους επιχειρήματα και τις δικές τους αξίες. Δύο παραδείγματα να σας δώσω για το πώς ε, αφαίρεσε άτομα από τα δίκτυα της ίσης ένα άτομο από τη Φιλανδία. Όχι τόσο μακριά από εσά. Ήταν ο υπαριθμόν 2 άγγλοφωνος ε, λογαριασμός του ίσης. Ενάμιση, άτο... χρόνο πέρασα με το άτομο αυτό του. Μιλούσα πάρα πολύ όμορφα. Τον, ε, προσπάθησα να τον πείσω με παραδείγματα από το Κοράνι. Μιλούσαμε. Ακόμα και φιλία μπορώ να σας πω ότι σας ε, πω ότι του έδωσα. Και έφυγε λοιπόν από το δίκτυο αυτό και τώρα έχει στραφεί εναντίον του. Είναι κατά του ίσης, κατά του Ισλαμικού κράτους, κατά του εξτρεμισμού και ε, ενεργοποιείται. Χρησιμοποιώ λοιπόν τον ίδιο μηχανισμό προσελτισμού ουσιαστικά που χρησιμοποιεί το Ισλαμικό κράτος κατά του Ισλαμικού κράτους. Δηλαδή μιλάω στους νέους, τους εξηγώ τις ε, και τότε ο νέος αυτός είναι αυτή ενδεχομένως να επιχειρηματολογούν με τον ίδιο τρόπο. Ε, ένα άλλο κορίτσι, λευκό, από τις ΙΠΑ, προσπαθούσαν να την ε, να χρησιμοποιήσουν ε, μέσω Twitter, μέσω tagging, μέσω μηνυμάτων και ευτυχώς και αυτή σταμάτησε και δεν μετέβησε στη Συρία. Έχω κάποιες ε, ιστορίες, ε, επιτυχίες τέτοιες, αλλά υπήρχαν και αποτυχίες ασφαλώς. Δεν μπορεί να τους σώσουμε όλους. Για κάποιους νέους, πολύ απλά αυτή είναι η κατεύθυνση που θα πάρουν στη ζωή τους. Στο σημείο 3, το πώς μπορούμε να τα θέσουμε όλα αυτά σε μια κλίμακα, στον ιδιωτικό κλάδο ε, δεν μπορεί να κάνει λεφτά η κυβέρνηση. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση να διευκολύνει τις συναντήσεις μεταξύ ΜΚΙΟ και ιδιωτικών ε, ε, ομίλων, ενώσεων που είναι δεδεθειμένες ε, να πληρώσουν, να δώσουν χρήματα, αλλά δεν κατανοούν απαραίτητα σε ποια μεθοδολογία θα πρέπει να επενδύσουν. Άρα θα καλέσω το Κοινοβούλιο, τους βουλευτές, ε, να το κάνουν αυτό, να διευκολύνουν και να οργανώσουν ε, συναντήσεις μεταξύ προσώπων της ε, μουσουλμανικής κοινότητας και ε, μεταξύ άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν εντάξει δει ότι έχετε χριστιανούς, Εβραίους, ακόμα και ε, άθεους που θέλουν να ζήσουν όλοι στο ίδιο περιβάλλον, όταν λοιπόν κινητοποιηθούν όλες αυτές οι φωνές, όλα αυτά θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από μία μόνο Ισλαμική, μουσουλμανική φωνή στο ίντερνετ που λέει ότι όχι το Κοράνι λέει αυτό. Σε ό,τι αφορά τις μεγαλύτερες προκλήσεις, ε, για να συνεχίσω από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενοι μελητές, είναι η ρωσική προπαγάνδα και η χρήση των ιστοριών κατά των μεταναστών. Και υπάρχουν ε, διάφορα ε, ρωσικά στοιχεία. Υπάρχουν και Γάλλοι πολιτικοί που ζητούν ε, χρηματοδότηση της πολιτικής της εξωτερίας από τη Ρωσία. Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις και θα δημιουργήσουν ένα δεύτερο επίπεδο ανησυχίων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και για την αστυνομία και για τις δικές υπηρεσίες. Γιατί αφενός θα πρέπει να παρακολουθούν τα μέλη της ΔΑΕΣ, κατά δεύτερον θα πρέπει να παρακολουθούν τις μεταναστευτικές ροές Και όχι μόνο κατά πόσον υπάρχουν ε, μαχητές ανάμεσα στους ε, πρόσφυγες ή αν οι πρόσφυγες που δεν είναι ριζοσπαθικοποιημένοι παρακολουθούν ε, τα μηνύματα κατά των μεταναστών, αυτό ενδεχομένως να τους οδηγήσει σε ριζοσπαθικοποίηση και κατά τρίτον τη βία κατά των μεταναστών. Χάρηκα ιδιαίτερω που στις Βρυξέλλες πριν από κάποιες ημέρε είδα ότι κάνατε ένα ράλι κατά του μίσου όπου εμφανίστηκαν εκατοντάδε ε, άνθρωποι. Αυτά πραγματικά ακούγονται και αυτά είναι μηνύματα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουν, να συνεχίσουν να δίνονται. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι όσο πιο πολύ το καθεστώς σα κάλυπτε διπλωματικά χθες μόλις ε, ε, χτύπησαν με βόμβες και προκάλεσαν θάνατο δεκάδων ε, ανθρώπων. Όσο πιο πολύ λοιπόν διατηρηθεί το καθεστώς Ασάντ, τόσο πιο πολύ θα έχει η ουσία υπόσταση ε, το Ισλαμικό κράτος. Γιατί το Ισλαμικό κράτος βγαίνει και λέει ότι καταπολεμούμε το καθεστώς του Ασάντ, το καθεστώς του Ασάντ λέει ότι θα πρέπει να μας υποστηρίξετε εμά γιατί ή εμείς θα επικρατήσουμε οι τρομοκράτες, αλλά η ουσία είναι ότι ο Ασάντ είναι ο τρομοκράτης στη Συρία έχει πολύ πιο πολύ εμπειρία, πολύ πιο πολλά χρόνια εμπειρία στο βασανισμό, βιασμό και στις δολοφονίες ανθρώπους. Αν δεν αντιμετωπιστεί λοιπόν το σημείο αυτό, η τάση θα αποτελεί σύμπτωμα απλό ενός μεγαλύτερου προβλήματος και θα προσπαθούμε να το επιλύσουμε, αλλά δεν θα καταφέρνουμε να το επιλύσουμε. Κλείνοντας, σε ό,τι αφορά την επιστροφή των αλλαδαπών μαχητών, η χρήση των πρώην εξτρεμιστών είναι μια πάρα πολύ ωφέλιμη ε, προσέγγιση και αυτό θα πρέπει να το βρουν ως λύση οι μυστικές υπηρεσίες. Πώς ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιες πρακτικές. Δεν μιλάω για άτομα που επιστρέφονται ε, από, την, από το Ισλαμικό κράτος. Μιλάω για άτομα που έχουν φύγει πριν από πάρα πολλά χρόνια και είναι παραγωγικοί στην οικογένεια, στην κοινωνία και μπορούν να παρουσιαστούν ως επικοδομητικά μέλη της κοινωνίας. Αν ένας αγαταπός λοιπόν μαχητής ε, ζητά να ξαναμπεί στη χώρα σας, θα πρέπει να το κάνετε, θα έλεγα, προϋπόθεση να βγουν δημόσια και να προβάλλουν τα μηνύματά τους. Γιατί οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. έχω συνεργαστεί στενά με κυβερνήσεις, μπορούν να στραφούν ε, στον τομέα της ε, πρόθεσης μηνυμάτων και της ασφάλειας και έχουν το ρόλο τους να διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις και οι ΜΚΟ έχουν μεγάλο ρόλο να διαδραματίσουν για να κινητοποιηθεί λοιπόν ο κόσμος αυτός ο οποίος τα έχει κάνει αυτά στο παρελθόν αυτό θα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την, ε, τα μηνύματα της ΝΤΑΕΣ. Σας ευχαριστώ πολύ σε ευχαριστώ. Και τώρα θα συζητήσουμε. Ο μιλητέ είναι πολύ ομάδα, Κύριε Σουγκουριάνο. Okay, thank you very much. Uh, ευχαριστώ πολύ. Στις ερωτήσεις θέλω να πάω. Θέλω κάποιες διευκρινήσεις Άκουσα τον κύριο Ρέντμαν. Ανέφερε την Daily Mail και την εκστρατεία της. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κάνει περίπου τα ίδια πράγματα. Δεν έχει σημασία ότι κάνουν εκστρατεία για το σωστό. Αν δείτε την εκστρατεία για το να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει η κυβέρνηση βλέπετε την ίδια διαφθορά και πειραγμένα στατιστικά κλπ. Δεν θα περιόριζε αυτού του είδου την εκστρατεία σε ένα στατόπεδο ή σε άλλο στατόπεδο. Δυστυχώ, συμπεραίνω ότι και τα δύο στατόπεδα όσον αφορά το βρετανικό δημοψήφισμα διαπράττουν το ίδιο έγκλημα. Τώρα για τις λύσεις είχα την εντύπωση ότι θα πρέπει να εφεύρουμε ή να επανεφεύρουμε τα ΜΜΕ, αλλά έχουμε τα μέσα ενημέρωση. Ερώτηση. Ένα κομμάτι του προβλήματος Μήπω οφείλεται στο εξή. Τα επικρατώντα μέσα ενημέρωσης, την, ε, μάλλον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ δεν ε, λένε πάντα την αλήθεια, δεν κατονομάζουν πάντα. Καμιά φορά διστάζουν να μιλήσουν, να πούν την αλήθεια, πολλά ε, θέματα δεν προβάλλονται αρκετά ή δεν αναφέρονται καν. Όσον αφορά τη Ρωσία, Φερρυπίν. Πολλές από τις ειδήσει που αφορούν τη Ρωσία είναι εκεί διότι ο πρόεδρος Πούτιν είπε ή δεν είπε κάτι. Η κάλυψη για το Ισλαμικό κράτος δυστυχώς οφείλεται στην πορνογραφία της βίας όπως δυστυχώς μπορώ να την αποκαλέσω. Τέλος. Δεν αναφέρατε κάτι άλλο. Αφού μιλάμε για ρωσική προπαγάνδα και ότι υποβόσκει και χρησιμοποιεί έτσι κρυπτές διαδικασίες. Οι εξαγορές μη μη έψιλον διεκπροσώπων χρησιμοποιούνται ρωσικά χρήματα κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι πλέον αστείο αυτό. Ε, ποια είναι η άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Ο κ. Φράνκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω δηλώνοντας ότι ήμουν δημοσιογράφος επί 40 έτη. Και λυπούμε που έχασα τον συνάδελφό μου εκεί στο βήμα, διότι ο Μπροκ απεχώρησε. Είδα ότι ξεκίνησε τις παρατηρήσεις του κάνοντας παρομοίωση. Αναφέρθηκε στο Βιετνάμ. Ποιο ήταν το μάθημα του πολέμου στο Βιετνάμ και των ΜΜΕ. Θα έλεγα ότι επεκράτησε η αλήθεια. Τα ανεξάρτητα ΜΜΕ απεκάλυψαν φρικαλαιότητες που διαπράχθησαν από τις ΗΠΑ και μακροπρόθεσμα έδειξαν ότι αυτός ο πόλεμος δεν μπορούσε να κερδιθεί και ο πόλεμος του Βιετνάμ ελάμβανε χώρα σε εντελώς διαφορετικό τοπίο ΜΜΕ από το σημερινό. Ε, ε, λιγότερους αναγνώστες έχουμε, λιγότερους θεατές, λιγότερους... Δεν υπήρχαν τα κοινωνικά μέσα τότε. Οι ταινίες που γυριστήκαν για τον πόλεμο του Βιετνάμ έπρεπε να σταλούν πρώτα στην Ιαπωνία και να εκπαιμφθούν στις ΗΠΑ. Χρειαζόταν δύο μέρες για τα επίκαιρα να παρουσιαστούν στις ΗΠΑ. Πριν αποφασίσουμε με το τι πρέπει να κάνουμε στον περιπλοκότατο τομέα, πρέπει να δούμε ποια είναι η επιρροή της ρωσικής προπαγάνδας, αυτής της επίθεσης προπαγάνδας. Πόσος κόσμος παρακολουθεί τις ρωσικές ειδήσει τακτικά στις διάφορες χώρες. Στις χώρες που έχουν ρωσικά ΜΜΕ ή ρωσική α, μειονότητα στην οποία απευθύνονται την προπαγάνδα. Και το εξή ερώτημα μπορούμε να θέσουμε. Θέλουμε να αυξήσουμε τον ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία και σε άλλο μέτωπο, στα ΜΜΕ. Ο κ. Ρέντμαν είπε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους το δημοψήφισμα στην Ολλανδία χάθηκε για την ευρωπαϊκή πλευρά ήταν διότι είχαμε ρωσική προπαγάνδα και την άκουσε ο λαός. Δεν χρειάζομαι ρωσική προπαγάνδα για να καταλάβω ότι η Ουκρανία πράγματι είναι διεφθαρμένη χώρα. Αυτό κάθε φορά το λέει σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ρωσική προπαγάνδα. Δυστυχώς είναι γεγονός. Και ήταν αλήθεια επί σειρά Τέλος. Να ρίξουμε και το φως σε παρόμοια προσπάθεια. Το Al Jazeera USA. Άλλη προσπάθεια. Με μεγάλες προσδοκίες ξεκίνησε αυτό το κανάλι και ξέπεμψε στις 30 Αυγούστου του 2013. Αποστολή του μεταξύ άλλων ήταν να παρουσιάζει αντικειμενική άποψη για τον αραβικό κόσμο, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και να ρίξει διαφορετικό φως για τα γεγονότα στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε 11 μέρες, στις 30 Απριλίου, θα κλείσει το Αλτζαζίρα αυτό. Εκατομμύρια ε, δολάρια χάθηκαν και πολλά ταλέντα θα πρέπει να, να συγγνώμη, να προσέχουμε γιατί πράγμα ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Ο κ. Ολτροβίτσιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να πω ότι ξεκινήσαμε ενδελεχείς συζητήσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την προπαγάνδα, για την πλήση εγκεφάλου και για τους πολέμους πληροφόρησης που λαμβάνουν χώρα γύρω μας. Έπρεπε να φτάσουμε αυτό το σημείο πολύ πιο πριν, όχι τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ Γι' αυτό θα πει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από την έξι σχέση φορτίγα να βγάλουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Κυρίως όσον αφορά τα πρακτικά αποτελέσματα. Έχουμε την κοινωνία της πληροφορίας και ο καθένας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες επιθυμεί. Δύσκολο να υπάρχουν κεντρικές πηγές που να επιβάλλουν κάποιες απόψεις. Οι άνθρωποι είναι πιο ελεύθεροι. Έχουν καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και στην έρευνα για τις πληροφορίες βάσει κριτηρίων. Αυτή η συζήτηση μας οδηγεί σε κάτι καινούριο. Σε κάτι από το οποίο μπορούμε να αποφεληθούμε, εάν λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταλάβουμε το εξή ότι ο πόλεμος των πληροφοριών και η πλήση εγκεφάλου χρονικώς πώς διαφέρουν. Δεν προξενούν φυσική ζημία. Ο χρόνος που δαπανάτε για για ζημιά που προκαλείται στον κόσμο επιβάλλοντας κάποια πλαίσια σκέψεως. Δεν αλλάζει τον κόσμο τόσο γρήγορα, γιατί ο κόσμος χρειάζεται χρόνο να αλλάξει τρόπο ζωής και νοτροπία. Σημειώνω αυτά που είπαν τα μέλη του πάνελ. Είναι κάτι που αφορά την αλληλουχία γενναιών, Άρα δεν είμαι αισιόδοξο για την ρωσική κοινωνία. Η κοινωνία μετά τον Πούτιν δεν θα μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Η πλήση εγκεφάλου θα αφήσει ίχνη. μακρόν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ερώτηση προς όλα τα μέλη του πάνελ τροφή προς σκέψη. Κυρίως αυτό φορά τον Καναδό συνάδελφο. Αν συγκρίνουμε τον Τάις, το Ισλαμικό κράτος και τη ρωσική προπαγάνδα, πώς δυσδύουν στην ε, Αμερικανική κοινωνία, ποια προπαγάνδα είναι πιο επιτυχής. Κάνω συγκρίσεις. Είναι πολύ επιθετική η προπαγάνδα τους. Επιδιώκει στόχους. Δεν είναι καθόλου αθώα προπαγάνδα. Θα συνέκρινα τις δύο προσπάθειες. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο επικίνδυνη. Και οι δύο βασίζονται στην ιδεολογία. Κάποια ιδεολογία. Η ρωσική προπαγάνδα βασίζεται σε κρατική ιδεολογία. Είναι καλοπληρωμένη, καλοσυντηρούμενη, με πολλούς πόρους κάθε μορφής και πολιτικούς πόρους. Διερωτώ με όμως, ποια είναι η πιο επιζήμια για την κοινωνία, κυρίως τον είπα, προς τους Ευρωπαίους, τα ευρωπαϊκά μέλη του πάνελ. Έχω μια ερώτηση. Για πρακτικές αποφάσεις. Σωστά αναφέρθηκε ότι η οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα ίσως θα πρέπει να τροποποιηθεί, να είναι στόχος μας. Μπορείτε να διευκρινίσετε. Τι είναι η τρόπο τι συστήνετε. Πώς θα αλλάξει την οδηγία. Πώς θα το κάνατε αν είχα την εξουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στουρβούτσιος. Και τώρα θα μιλήσω εγώ με τη σειρά μου. Είμαι βουλευτής της ε, Ενωμένης Αριστεράς στην Ισπανία και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Αριστεράς. Νομίζω ότι όλα αυτά σαν προπαγάνδα αντιρωσική ήταν τέλεια και οπότε βρήκαμε μια κλασική ωραία, ωραίο ορισμό της προπαγάνδας. Ε, μανιχαϊσμός, ε, υπεραπλούστευση, το απόλυτο κακό και όλα αυτά με στρατιωτικό λεξιλόγιο. Έτσι τα είπαμε. Ακριβώ όπω γινόταν και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εξαρτάται και αυτό από το πώ το βλέπει κανείς το θέμα. Τι δεν έκαναν όμω τον πόλεμο του Ιράκ, είπα, δεν παραπληροφόρησαν, δεν είπαν ψέματα, δεν δημιούργησαν δίθεν πηγές, δεν θύμωσαν τους δημοσιογράφου που δεν τους άρεσαν. Να, ένα κλασικό παράδειγμα προπαγάνδας, τον είπα που την πετάξανε σε όλο τον κόσμο. Και έτσι αποσταθεροποίησαν ουσιαστικά όλη τη Μέση Ανατολή. Και να μην μιλήσουμε για τον πόλεμο τέταρτης γενιάς όπως ε, λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Δηλαδή ψυχολογικό πόλεμο, δίκτυα και πόλεμο μέσα από την κοινωνία των πολιτών. Για να δούμε μιλάμε για ασφάλεια και λένε για την ε, Ουκρανία, μιλούν για φορητούς φούρνους. Αυτό δεν είναι προπαγάνδα. Ή λένε για την προπαγάνδα της συμμαχίας κατά της Ντάις που έχουμε 60 χώρες που επί ένα έτος και παραπάνω βομβάρδιζαν τους τρομοκράτες του Ντάις και δεν προχώρησαν ούτε μία σπιθαμία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προσβλητικό το να συγκρίνει κανεί το Ισλαμικό κράτο με τη Ρωσία. Διότι ανήκει στο ΝΟΙΕ, είναι ένα κράτο η Ρωσία και σέβεται τι σχέσει τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να την συγκρίνουμε με τους ε, τρομοκράτες που κόβουν λαρίγια και που σκοτώνουν κόσμο και εξοντώνουν μειονότητες. Όταν εγώ δουλεύα σε μιλούσαμε για αυτές τις εκτελέσεις χωρίς δίκη αλλά το θέμα είναι τις τρίτες και τετάρτες στο βάλε γραφείο του Λευκού Οίκου πώς αποφασίζουν για τις ε, εκτελέσεις τις εξοδαφικές και χωρίς δίκη που κάνουν με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Να ο μανιχαϊσμός. Για μένα στην Ουκρανία είχαμε ένα πραξικόπημα και ξέρουμε όλοι ποιοι τα έκαναν αυτά. Ξέρω πολύ κόσμο που το πιστεύει αυτό. Εγώ τι να σας πω. Ε, να, έχουμε ας πούμε και την επιχείρηση Κόσοβο. Μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια τεχνητή χώρα, τεχνικό κράτος. Εκεί που είναι όλοι λαθρέμποροι, έμποροι όπλων και κάνουν και εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Τα είδε αυτά η Κάρλο Πόντε, η οποία μια που δουλεύει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ε, αυτό πάνε να πει ότι είναι Ρωσίδα, έτσι δεν είναι. Να δούμε τώρα πώς βλέπει ένας δημοσιογράφος για όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση ΜΜΕ σε λίγα χέρια, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες αντισταθμίσεις, θα πρέπει να υπάρχει πολυφωνία και ελεύθερη επιλογή από πλευρά του κόσμου. Είπαμε για το Russia Today και Και δεν είναι σωστό αυτό που μιλήσατε για τα ΜΜΕ, αλλά μιλήσατε με όρου στρατιωτικού. Κύριε Σάφχα, ζωήτε το λόγο. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για αυτά που είπε, τα οποία εγκρίνω προφανώ. Δεν είναι συχνό να έχουμε έναν Πρόεδρο που είναι κάπως ανατρεπτικός ε, λέγοντας την αλήθεια. Πάνω σε αυτά που είπατε, να σας πω ότι είμαι συνηθισμένος στην προπαγάνδα. Αλλά έχουμε συνόδους... Φτάσαμε τα όρια, τα νότατα της προπαγάνδας. Κύριε Ράιτμαν, ενώπατη της δημοκρατίας. Να σας περιγράψω τη δική σας λογική. Εν ονόματι της δημοκρατίας ξεκινάτε λέγοντας ότι είσαστε αντίθετο στο δημοψήφισμα. Ιδιαίτερα στο δημοψήφισμα στην Ολλανδία, στη Δανία και στη Γαλλία ενάντια στα δημοσιοφίσματα, ονόμα της δημοκρατίας. Λέτε κύριε Ρέντμαν της αντίθετο στο Ισραήλ, σαν τη μοναδική χώρα που είναι δημοκρατική, που έχει 20% Άραβες εντός του, των ορίων. Εν ονόμα της δημοκρατίας είστε αντίθετος λοιπόν ε, με το λαό και με τα συστήματα που επιτρέπουν τη λειτουργία της δημοκρατίας. Να ένα παράδειγμα προπαγάνδας. Δεύτερον, ψεύδος. Μιλάτε για δημοσκόπηση, για δημοσκοπήσεις, για την Κρυμαία. Έγινε δημοψήφισμα. Αμερικανικό την ε, διέπραξε τη δημοσκόπηση των Γκάλοπ. Υπενθυμίστε τα στοιχεία, να σας δώσω τις δημοσκοπήσεις αν θέλετε. Μετά, να πω και κάτι άλλο. Τι είναι η προπαγάνδα Επιτρέψτε μου να συνοψίσω προπαγάνδα. Δεν συμμερίζομαι αυτό που θα σας είπω, αλλά ειδού η προπαγάνδα. Είστε αντίθετο κατά τη δημοκρατία, μπορώ να πω ότι είστε φασίστα. Επειδή είσαστε κατά του Ισραήλ, μπορώ να πω ότι είστε αντισημίτης. Επειδή είστε υπέρ της προπαγάνδας, διότι δεν θέλετε να αναλύσετε τη δική σας προπαγάνδα και την καταγγέλλετε αυτή των άλλων, θα έλεγα ότι είσαστε ο επικατέστορος προπαγανδιστής. Λοιπόν, αν είστε πραγματικός προπαγανδιστής, είσαι φασίστης, αντι, ε, φασίστας, ε, αντισημίτης. Και φύρερ της προπαγάνδας. Ο κ. Σανόφσκι, να σας υπενθυμίσω ότι ο στρατηγός Ντεγόλ με το ΟΡΤΕΦ δημιούργησε, διόριζε τον επικεφαλής της, ε, της αλυσίδας. Ήταν, πιστεύετε, ότι ήταν φασίστας αυτός που έσωσε τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Γιατί θέλετε όταν τα ΜΜΕ είναι στα χέρια της αντιπολίτευσης ή στα χέρια ομίλου καπιταλιστικού που χειραγωγείται από ολιγαρχία, γιατί θέλετε να είναι πιο δημοκρατικό αυτό, γιατί θε... θεωρείται αυτή η προπαγάνδα είναι καλύτερη από αυτή που συντηρεί μια νόμη κυβέρνηση που έχει δικαίωμα να ειναι πιο δημοκρατικο αυτο γιατι θεωρειται αυτη η προπαγανδα ειναι καλυτερη απο αυτη που συντηρει μια νομιμη κυβερνηση που εχει δικαιωμα να εκφρασει την άποψή της με εψιλον τουλάχιστον που αντικατοπτεί στην άποψή τη. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Πολωνία. Τώρα, όσον αφορά τις κατηγορίες ε, κατά της Ρωσίας, μπορώ να μιλήσω για του Αμερικανού που έχουν περισσότερα μέσα που κάνουν προπαγάνδα. Όσον αφορά το παρελθόν και όπω δημιουργούν του μύθου του παρελθόντο. Θα μπορούσαμε να για τους cowboys και για τι αμερικανικέ ταινίε που δείχνουν το μεγαλείο της Αμερικής που πάντα νικάει. Και όσον αφορά την ασφάλεια θα μπορούσα να σας μιλήσω όταν μιλάτε για τα προβλήματα της ασφαλείας, για το ΝΑΤΟ και για τις εντάσεις που οδηγούν που υπάρχουν στον οργανισμό και καθοδηγούν τον οργανισμό. Ο κ. Μπρέτλοφ στην ομιλία του ανεφέρθηκε σε πολέμους και τάσει. Όλα αυτά δεν είναι πολύ σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά. Τώρα, όσον αφορά την πρακτική του, της τρομοκρατίας ε, με το έμβημα το μουσουλμανικό. Συμφωνώ μαζί σας, δεν πρέπει να αναμειγνύουμε τα πράγματα. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει φονταματαλισμός μουσουλμανικός που στηρίζεται στην Αραβική, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στους αδελφούς μουσουλμάνους. Ποιος τους υποστηρίζει. Ε, δεν, είχα, δεν κάναμε λάθος εμείς οι Δύσοι να συμμαχίσουμε με εκείνους που σπρώχνουν προς εξτρεμιστικά οράματα και φονταμελιστικά οράματα για το Ισλάμ. Και όταν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Ισλάμ και Ισλαμισμού, κάποιος Γάλλος που οφείλει στον Σαλ Μαρτέλ ε, που έδιωξε τους ε, Άραβες και που παντού όπου υπάρχει πλειοψηφία χριστιανική έχει εκριζωθεί από το Ισλάμ διότι αυτό είναι πραγματικότητα είμαι και τότε θεολόγος και είμαι ιστορικός των θρησκειών πώς θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχει η ανοχή εντός του συστήματος, διότι εγώ βλέπω ότι πραγματικά γίνεται. Τούτου λεχθέντος πιστεύω ότι κάναμε λάθος και κλείνω όσον αφορά τη σύγχυση που δημιουργήσατε. Το υπογράμμισε ο πρόεδρος μεταξύ ε, Ρωσίας και Ντάες. Εκεί ξεπεράσατε όλα τα όρια που μπορούν να ξεπεραστούν. Η ντροπή δεν σας συγκράτησε, δεν ντραπήκατε όταν φτάσατε σε τέτοιες υπερβολές και υπερβάσεις. Σας ευχαριστώ. Αυτά που είπατε και οι τρεις είναι σκανδαλώδη και δεν θα άξιζαν να ακούσαν να ακουστούν σε αυτό το κοινοβούλιο αν είχε ακόμα το συνέστημα της δημοκρατίας του λαού, το κοινοβούλιο και του κοινού καλού. Ευχαριστώ. Ξεκαθαρίζω ότι πριν μίλησα όχι βεβαίω ως πρόεδρος, αλλά ως βουλευτής, γιατί ο πρόεδρος έχει θεσμικό ρόλο και πρέπει να εξασφαλίσει όλοι να λαμβάνουν το λόγο. Μίλησαν όλες οι πολιτικές ομάδες και τώρα οι βουλευτέ τρία λεπτά. Ο καθένα κύριε Πιτίδη, έχετε το λόγο. Τρία λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όπω γνωρίζετε, η προπαγάνδα είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα, όχι μόνο από κράτη, όχι μόνο από εμπολέμου, αλλά και από οργανωμένε ομάδε ανθρώπων ε, και από ανθρώπου οι οποίοι ήθελαν να εξυπηρετήσουν διάφορα συμφέροντα. Ε, στη σημερινή εποχή η προπαγάνδα ε, έχει εξελιχθεί σε πραγματική επιστήμη. Άλλωστε, α μην ξεχνάμε ότι ακόμη και οι διαφημίσει είναι μια μορφή προπαγάνδα. Στι δημοκρατικέ ε, χώρε η αντιμετώπιση τη προπαγάνδα είναι δύσκολη διότι υπάρχει ελευθερία λόγου, υπάρχει δυνατότητα προσβάσεω σε πολλά μέσα. Άρα λοιπόν κάποιο που θέλει να προσβάλλει τα, ε, την κοινωνία την ευρωπαϊκή είναι πολύ εύκολο να το κάνει. Όμω μπορούμε να προστατεύσουμε, μπορούμε να θωρακίσουμε του λαού και τι κοινωνίε μα κατά της προπαγάνδας από όπου και αν προέρχεται αυτή υπό την προϋπόθεση θα εφαρμόσουμε κάποιες αρχές και κάποιες τακτικές. Η πρώτη και βασική αρχή είναι ότι πρέπει να, κάθε κράτος να λέει στο λαό του την αλήθεια. Και όταν λέω αλήθεια εννοώ να μην γίνεται το ίδιο το κράτος προπαγανδιστής και να παρουσιάζει είτε απόψεις που το εξυπηρετούν είτε απόψεις οργανωμένων ομάδων πιέσεως και διαφόρων συμφερόντων αυτή η τακτική μπορεί να ε, έχει επιτυχία σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Δεν μπορεί όμως να έχει ε, επιτυχία σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου ο κόσμος μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ποιο είναι το αληθές και ποιο είναι το ψέμα. Έπειτα μια βασική αρχή της προπαγάνδας είναι να υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ των όσων λέει και των όσων πραγματικά συμβαίνουν. Άλλο ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η μη δαιμονοποίηση του αντιπάλου μας. Δεν μπορεί δηλαδή να αποδίδουμε στον οποιοδήποτε αντίπαλό μα το απόλυτο κακό. Στη σημερινή εποχή βλέπουμε ότι μια τέτοια προσπάθεια γίνεται με τη Ρωσία, με τον Πούτιν, γίνεται με τον Άσαντ στη Συρία, όπου αυτή είναι το υπέρτατο ε, κακό και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι καλοί, είναι οι άγγελοι. Μια τέτοια προσέγγιση είναι δεδομένο ότι είναι θνησιγενής. Θα αποτύχει εξ αρχής, διότι πλέον ο κόσμος δεν είναι ανόητο, ούτε έχει δεν έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται. Άρα λοιπόν μια τέτοια προσπάθεια θα πέσει στο κενό και θα γίνει αναξιόπιστο το κράτος. Άλλο ένα αντίστοιχο στοιχείο είναι ότι δεν πρέπει να υπερτιμούμε τον οποιοδήποτε αντίπαλό μας. Κάτι το οποίο συμβαίνει δυστυχώς με τους τρομοκράτες του ISIS. Βλέπετε οι εικόνες είναι πολύ δυνατές συναισθηματικά. Βλέπουμε ανθρώπους να σφαγιάζονται από τον ISIS βλέπουμε να κάνει διάφορες τρομοκρατικές ε, δραστηριότητες και αυτές φοβίζουν τον κόσμο, άρα δίνουμε την δυνατότητα στην προπαγάνδα να υπερτιμήσει αυτόν τον αντίπαλο. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα δικά του πιστεύω και ποια είναι η δική του προπαγάνδα. Έτσι λοιπόν θα ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο. Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον κόσμο μας με αγάπη και συμπάθεια, να διαπαιδαγωγούμε σωστά και να μην στρεφόμαστε εναντίον του. Παράδειγμα χάρη, όταν δημιουργούμε ανεργία στους νέους, όταν παίρνουμε τα σπίτια από τον κόσμο, όταν του κλέβουμε ουσιαστικά την περιουσία, όταν τον γετοποιούμε ή τον απομονώνουμε, τότε δεν μπορούμε να, να ελπίζουμε ότι η εχθρική προπαγάνδα δεν θα έχει επιτυχία στη δική μας κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Gracias. Όλα την έχει το λόγο. σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ μα για το γεγονό ότι μοιράστηκαν μαζί μα τις ε, χρήσιμες, τη χρήσιμη εμπειρία του, Εδώ και πολλά, μάλλον πολλά χρόνια ε, έζησα υπό το καθεστώς ρωσική προπαγάνδα, στη Σοβιετική Ένωση, τη Σοβιετική Προπαγάνδα. Για να είμαι ειλικρινή, λοιπόν, οι τεχνικέ και οι τακτικέ ήταν οι ίδιε διαστρέβλωση της αλήθειας, χειραγώγηση της δημόσιας και κοινής γνώμης. Τώρα όμως έχουμε ένα νέο πεδίο εφαρμογή για την εφαρμογή της προπαγάνδας στα κοινωνικά μίντια. Τεχνικές που μπορούν να αγγίξουν τους πάντες. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο λοιπόν. Ένα ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι το εξή. Η ποιότητα της δημόσιου διαλόγου σε ό,τι αφορά την αλήθεια, σε ό,τι αφορά την προσδοκία του κόσμου για την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο τομέα. Γιατί όπως ακούσαμε μόλις, ο διάλογος αντικαθιστάται από τα συναισθήματα της ε, προπαγάνδας, που προκαλεί η προπαγάνδα. Και όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, οι Ντάε και τα θύματα της ε, έχουν εκτεθεί στην κοινή γνώμη. Τα θέματα του Ασάντα όμως που είναι πολύ πιο πολύ άριθμα δεν τα γνωρίζουμε. Και αυτό έχει συναισθηματική διαφορά, Βάρο σε ό,τι αφορά τη συναισθηματική ε, διαφορά σε ό,τι αφορά το συναισθηματικό βάρος. Άρα θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αλήθεια, γιατί είναι σημαντικό αυτό, η αλήθεια είναι αυτή που μας ε, κάνει δυνατού. Αλλά σήμερα επικρατεί η άποψη ότι η αλήθεια είναι σχετική και ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές αλήθειες. Να παρουσιάσω κάποιες ιδέες από αυτές που παρουσιάζονται. Σε ό,τι αφορά τους αντιπροσώπους, ο πόλεμος με τους αντιπροσώπων. Ε, οι εμπειρογνώμονες, η στήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Μιλώντας για τη Ρωσία, ξέρουμε την εφημερίδα που διατίθεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμα. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να είμαστε άμεση και να εξηγούμε τις αξίες μας. Ποιες είναι οι αξίες μας, είναι τρόπο ζωής μας ή κάτι πιο βαθύ. Κάτι που έχει πιο πολύ συνέχεια. Και ένα ερώτημα που ήθελα να θέσω σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη συνέργεια μεταξύ των επιθετικών, αρνητικών μορφών προπαγάνδας, γιατί αναφέρθηκαν εδώ και κινούνται στα κοινωνικά μέσα μπορούν να αυξήσουν τον αντίκτυπό τους μέσω συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Κέλλαν. Ο επόμενος, ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ πρόεδρε και καλωσορίζω πάρα πολύ τη συζήτηση που γίνεται. Χρειάζεται, χρειάζεται και μη σας πω ότι έχει καθυστερήσει κιόλα. Γιατί αυτό που βλέπουμε στη συγκεκριμένη φάση είναι το εξή. Όντω βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολέμου όπου και τα μέσα ενημέρωση συμμετέχουν στον ευρετικό πόλεμο. Είτε μα αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρωτού όμως ε, στραφώ προ τι ε, σύντομε ερωτήσει μου, θα ήθελα να πω το εξή. Θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια διαδικασία όπου διάφοροι φορεί, όπω η Ρωσία, όπω το Ισλαμικό κράτο, οικοδομούν μέσα στην κοινωνία μας ένα πέμπτο πυλώνα, μέσα στα κράτη-μέλη μας με τον σκοπό να αποδυναμώσουν, να εξαλείψουν την ομόνια της έννοιας, της ένωσης. Να καταστρέψουν τις ιατρατικές ε, σκέψεις, σχέσεις, προκειμένου απομονωμένοι και απογοητευμένοι να μπορέσουμε να, να μπορέσουν να μας ε, υποτάξουν. Και θα ήθελα να πω το ίδιο για τον Τσάμπερλεν μετά την συμφωνία του Μονάχου. Να μην ξεχνάμε ποτέ τι είπε για τον Τσάμπερλεν και για την ψευδέστηση ότι με τα μέτρα συμφιλίωση η Ευρώπη θα μπορούσε να σωθεί, θα μπορούσε να προστατευτεί. Γιατί στην πραγματικότητα η συμφωνία του Μονάχου προετοίμασε απλά τους Γερμανούς Ναζί για να γίνουν αυτό που έγιναν και για να σχηματίσουν μια γιγαντία συμμαχία με γιγαντιαίο αντίκτυπο για την ανθρωπότητα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, όταν μιλάμε για την ε, Ρωσία, όταν μιλάμε για το Ισλαμικό κράτος, λοιπόν, θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη αυτά. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές ε, ομοιότητες στο σημείο αυτό. Τρει ερωτήσει να κάνω. Καταρχάς, πώς μπορούμε να ποινικοποιήσουμε τα website, τις ιστοσελίδες που κάνουν ε, ριζοσπαστικοποίηση και μέσω των οποίων στρατολογούν. Σημαντική συζήτηση γίνεται και στη Γαλλία. Τι μπορούμε να κάνουμε από νομικής άποψης για να καταπολεμήσουμε αυτούς τους ε, μηχανισμούς. Κατά δεύτερον, ποιος είναι ο ρόλος των ε, των ημάμιδων που αυτό ανακηρύσσονται οι ημάμιδες ξέροντας ότι είναι ιδιαίτερη σημασία τους στις κοινωνίες μας και τρίτον τι γίνεται με τη χρηματοδότηση χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωση, πολιτικών κομμάτων, ΜΚΟ, πολιτικών κομμάτων Γνωρίζοντα ότι ακριβώ ο σκοπό του είναι αυτό ο πέμπτος πυλώνας, προκειμένου να ριζώσει. Ο κ. Πανθέρη. Δύο σύντομες παρατηρήσεις και μια ερώτηση. Πρώτα όλα Δεν άκουσα τη συζήτηση, αλλά, αλλά από ό,τι κατάλαβα από την ανάλυση που που έγινε και προσπαθώ αυτά να τα συγκεράσω. Έχουμε προπαγάνδα με διαφήμιση. Υπάρχουν αυτών του δύο ειδών ε, προσπάθειες επικοινωνίας. Στην πολιτική έχουμε πρώτα πρώτα την προπαγάνδα από κάποια καθεστώτα που σήμερα γίνεται με κάποιες στατικές επικοινωνίας και με τη διαφήμιση διαφημίζεται ένα πολιτικό προϊόν. Και αυτό που θέλω να καταλάβω είναι θα πρέπει να εμβαθύνουμε, να διερευνήσουμε τη σχέση της διαφήμισης με την προπαγάνδα. Χαμογέλος τον έξω αυτά που συζητούσαμε γιατί η χειραγώγηση και η στρέβλωση της νοοτροπίας, της συμπεριφοράς των άλλων γίνεται από κάποια καθεστώτα και μεταξύ άλλων και ο Πλάτωνας είχε επισημάνει το πώς χειραγωγείται και μια γενική συνέλευση από κάποιες αγορεύσεις και έχει κάνει τη διάκριση του καλού από το αληθές. Αυτά όλα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και τώρα. Θα ήθελα να καταλάβω εμείς πού θα βρούμε αντίδοτα και κυρίως στις σύγχρονες κοινωνίες τι θα κάνουμε με αυτή την προπαγάνδα. Έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο για να μπορούσαμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της προπαγάνδας που απολύτω και της προπαγάνδας που πιάνει τόπο. Άρα θα πρέπει κανείς να αναπτύξει κρίση. Αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε. Την δυνατότητα του κόσμου να κάνει την διάκριση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλιώς κυριαρχείται κάποιος από τους φορείς της προπαγάνδας. Εδώ θα ήθελα να μου κάνετε μια διευκρίνηση. Σε ευχαριστώ. Και τώρα έχει ένα πεντάλεπτο ο κάθε ομιλητή τον οποίο δώσουμε το λόγο να γίνει μια σύνθεση ακριβώ με τη σειρά που μιλήσατε προηγουμένως. Κύριε Ρέτμαν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου ξαναδίνετε το λόγο. Μάλιστα. Εδώ κάπου δεξιά αναφέρθηκε το Brexit και οι σχετικές ε, εκστρατείες προεκλογικές. Ανησυχεί η κυβέρνηση για ε, τις οικονομικές συνέπειες. Δεν νομίζω ότι η εκστρατεία αυτή μπορεί να εξομοιωθεί με άλλες προσπάθειες όπως όταν είχαμε τις βόμβες εδώ τι είπε πριν πολύ πολιτική όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ ήταν κάτι κακό στα δημοσίευματα στο Daily Express και σε άλλες ταμπλόιτς Daily λέγανε ότι να, να την Ευρωπαϊκή Ένωση να τις βόμβες και βλέπουμε ότι υπήρχε επομένω ένα χαρμάνι ρητορική πολιτικής και ξενοφοβίας. Φωτογραφίες με τον κόσμο ε, να έχει χτυπηθεί από τις βόμβες και καμένος να τρέχει. Και βέβαια, να αυτό είναι, έτσι διαμορφώνεται η γνώμη από αυτούς τους spin doctors. Αν και δύο ομιλητέ επίση μα μίλησαν και για το Βιετνάμ. Και να δούμε τι γίνεται με τα Panama Leaks, τι γίνεται από πλευρά Ρωσία. Και έχουμε τις αποκαλύψεις για διαφθορά στο περιβάλλον το στενό του Πούτιν. Βέβαια θα λάμψει τελικά η αλήθεια, αλλά Είδατε τι έγινε με την προπαγάνδα επί πολέμου του Βιετνάμ στη ΣΥΠΑ. Ε, έκαναν τη δουλειά τους οι δημοσιογράφοι. Δεν φοβήθηκαν μήπως τους πυροβολήσουν. Κάποιος μίλησε για την πορνογραφία του Ισλαμικού κράτους, για την βία. Έχουμε πάρα πολλά κακά μέσα ενημέρωση. Σε αυτό θα μπορούσε να μας μιλήσει ο συνάδελφος από τον Καναδά. Πολύ βία μέσω μουσικής, μέσω παιχνιδιών κλπ. Και αυτό έχει επιπτώσει στους νέους. Κάποιο είπε ότι δεν χρειάζεται να μα πούνε οι Ρώσοι ότι είναι η Ουκρανία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όμω για κοιτάξτε πώ το πουλάνε αυτό οι Ρώσοι σε σχέση με το δημοψήφισμα. Ε, κυκλοφόρησαν πάρα πολλά ψέματα ότι θα γίνει μέλος η Ουκρανία για το πόσο αποτελεί η Ουκρανία ένα κίνδυνο για την ασφάλειά μας. Άρα το θέμα είναι το πώς παρουσιάζεται το πακέτο που πουλάει κανείς την προπαγάνδα. Όταν όμως πάμε στην οδηγία που λέει για τα κοινωνικά μέσα ενημέρωση και τη συνέργεια και πώς θα αντιμετωπίσουμε και την ριζοσπαστικοποίηση, ε, θα πρέπει να σας τα πούνε εδώ πέρα και οι παρακαθέντε τα ξέρουν καλύτερα, αλλά για την ζωσπαστικοποίηση έχω να πω ότι έχουμε την υποδομή ε, να καταπολεμήσουμε και την παιδική πορνογραφία σε συνεργασία με τη Microsoft και μεγάλες εταιρείες να συνεργαστούμε δηλαδή για την επιβολή του δικαίου. Από την άλλη μεριά, ε, πού είναι τα, όρια μεταξύ ε, εγκληματικής ζωσπαστικοποίησης και ζωσπαστικοποίησης ιδεολογικής όπως θρησκεία. Το θέμα είναι τι αποτελεί έγκλημα. Αν κάποιος έχει ένα website που λέει ότι πρέπει να γίνονται ανθρωποκτονίες στο όνομα του Ισλάμ, εντάξει. Όταν όμως ε, αυτό έχει να κάνει και με στρατολόγηση και λέει ότι πρόκειται να σας δώσουμε και λεφτά, θα σας φέρουμε σε επαφή με οργανώσεις, ε, τότε ένα τέτοιο site θα πρέπει να κλείνει. Ε, μου επιτέθηκαν φραστικά κάποιοι ομιλητέ όπως ο κύριος Σάφραζερ που έφυγε και είπε ότι ήταν προπαγανδιστής θα, θα με αποκαλούσε φασίστα και όμως να τον αποκαλέσω πολλά πράγματα αλλά λυπάμαι που έπαθε νευρική κρίση χειρότερα από τη δική μου τώρα που σας μίλαγε σας λυπάμαι τώρα για το κύριο ε, Περμούι εδώ ο πρόεδρος στα δεξιά μου είναι πολύ σημαντικό να καθιστούμε υπεύθυνε στις κυβερνήσεις Είδατε τι έγινε με τα Panama Leaks. Ε, βγήκε στο φως το σκάνδαλο και δεν υπήρξε επιλογή του ποιον θα προστατεύσουν οι δημοσιογραφοί και ποιον όχι. Κύριε Περμού, είναι αλήθεια ότι έχω διαφορετική πρόληψη από σας. Είμαι πολωνικής ε, καταγωγής και δραπέτεσαν από τον κομμουνισμό της οικογένεια μου, άρα έχουμε τελείως διαφορετικό παρελθόν και Λυπάμαι που κάποιο τόσο στρατευμένο και έξυπνο στον ίδιο περμό είπε ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση είναι κάτι σαν την κυβέρνηση του Πούτιν για την εξωτερική πολιτική. Είπατε ότι η αμερικάνικα μέσα είναι κάτι σαν το Σπούτινικ. Μα είπα προηγουμένω ότι αυκίνα τα μέσα εγκληματούν καλώντας η άσκηση βίας. Είναι το θέμα, υπάρχει αναχρονισμός, υπάρχει κακή ενημέρωση. Τίποτα δεν ωφελούν εκείνα τα μέσα ε, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της σήμερα. Ο κύριος Τζέσχη Πομενός και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Ζαν Λουίξ Αφχάουζερ. αποχωρήσατε. Δεν θα απαντήσω σε εκείνον. Θα εστιαστώ επί των άλλων ερωτήσεων που ετέθησαν. Έκανα σαφή διάκριση μεταξύ Ρωσίας, προπαγάνδας ρωσικής και Ντάες. Είπα ότι υπάρχουν ελάχιστα κοινά σημεία. Και ήθελα να πω ότι πρέπει να βρούμε ανάλογη αντίδραση, διαφορετικά μέσα και διαφορετική γλώσσα για την αντιμετώπιση αυτών. Αλλά επηρεάζουν εξίσου, μας επηρεάζουν εξίσου. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεύτερο ερώτημα αφορούσε πώς γίνεται εξαγορά μέσων ενημέρωσης με δια εκπροσώπων δια, ε, στην Ανατολική Ευρώπη. Το έφυξα αυτό. Έλεγα ότι είναι ένα από τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Να δούμε πού κρύπτονται οι, οι πόροι μέσω αντιπροσώπων προς επιχειρήσεις κλπ. που εξαγοράζουν ΜΜΕ και δεν αφορούν πραγματικό ανταγωνισμό στην αγορά. Είναι χρήματα που δίδονται για στρατηγικούς σκοπούς. Γι' αυτό ε, χρειάζεται προσοχή να δοθεί. Παράδειγμα, αφορούσε την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει εμπορικό κανάλι. Από τον Φιρτά στον Λιγάρχη που συνελήφθη στην Αυστρία. Το Ίντερ, το κανάλι αυτό, το μισό είναι στην κατοχή ε, ενός από τα βασικά ρωσικά κανάλια. Αν προσπαθήσετε να βρείτε στο διαδίκτυο τις πληροφορίες δεν είναι και τόσο εύκολο. Άρα, απάντηση να προσπαθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της οδηγίας για τα οπτικοκουστικά να πετήσουμε διαφάνεια όσον αφορά την χρηματοδότηση και την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης. Αυτό θα βοηθούσε. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε μέσω της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά. Αυτό μπορούμε να τη συνδέσουμε με την παρέμβαση του κυρίου Μποστινάρου. Πώς να κοπήσουμε στο σελίδας προσιλητισμού και στατολόγηση τους ριζοσπαστικούς ημάμιδες που προωθούνται μέσω του διαδικτύου και κανόνες για τη χρηματοδότηση των πυλών αυτών των διαδικτυακών και των σελίδων. Εγώ δεν είμαι ειδικό για την οδηγία περί οπτικοακουστικών. Όταν μιλώ με πυρογνώμονες αναφέρονται αυτοί σε σωστά εργαλεία για να αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ΜΜΕ ξεπερνάνε την κόκκινη γραμμή και κάνουν πράγματα κολάσιμα. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε σαφή διαχωριστική γραμμή αποδεκτού, μη αποδεκτού, νομίμου, παρανόμου. Αυτό θα βοηθούσε. Και θα μπορούσαμε από εκεί να συζητήσουμε πώς χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι πόροι που δίδονται στα ΜΜΕ για να εκτελέσουν αποστολή τους. Τώρα, αν υπήρχε πάντα ή όχι προπαγάνδα. Αυτό είναι εύκολο θέμα, πανεύκολο. Όταν μιλάνε οι άνθρωποι, οι μεν στους δεν προσπαθούν να επηρεάσουν ένα τον άλλο και στον κύριο Παντζέρη και σε πολλούς άλλους που το έθεσαν. Μόνο μια απάντηση υπάρχει και ένα φάρμακο. Ισορροπία στην πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης. Η ισορροπία άμα έχουμε ισορροπία επιλογές. Αν κανείς δεν με περιορίζει την επιλογή μου, μπορώ να επιλέξω σταθμό, όπως κάποιος θέλει να ακούσει ταυτόχρονα στο Sputnik και στο Fox. Εγώ δεν ακούω ούτε το Fox News ούτε το Sputnik. Όλοι μπορούν να διαλέξουν όμως τι θέλουν να ακούσουν. Θα πρέπει να έχουμε τις επιλογές. Αν πάμε στη Μόσχα, έχουμε περιορισμένες επιλογές. Και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα, όταν δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και επιλογές ο κ. Ζανλούκ Αφχάουζερ, αν θέλει να δημιουργήσει ένα κανάλι και να διορίσει το διευθυντή του καναλιού στη Μόσχα, σα διαβεβαιώνω ότι δεν θα πάει κάνει αυτό στη Μόσχα. Δεν είναι μια αγορά με δίκαιο ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των διαφόρων εμπλεκομένων. Τότε χαλάει η ισορροπία. Τότε δημιουργούνται ζητήματα. Και δεν μιλάμε για ένα φαινόμενο κοινό για την ανθρωπότητα τα τελευταία 2.500 χρόνια. Έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Ε, λυπάμαι δεν απάντησα σε όλες τις τεθείς ερωτήσεις που αφορούν τις δικές μου γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη μου. Σε άλλη περίσταση που ελπίζω να παρουσιαστούν και άλλες πολλές θα απαντήσω. Ευχαριστώ κύριε Κομιανόφσκι. Και τώρα... Ο κύριος έχει το λόγο για να απαντήσει. Νόμιζα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν ε, μάλλον βαρετό, αλλά δεν ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρώτο σημείο που αναφέρατε. Ήταν πάρα πολύ καλό το θέμα αυτό για τη συζήτηση κατά πόσον η ρωσική προπαγάνδα ή η προπαγάνδα της ΔΑΕΣ ε, είναι πιο επικίνδυνη. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε τους δεκάδες εκατομμύρια ε, μουσουλμάνους ε, που είναι στην Ευρώπη, 5.000 και κάτι από όλους αυτούς κατάφερε να στρατολογήσει η Ντάις. Αν τους συγκρίνουμε αυτούς με τους ανθρώπους που κινούνται προς τον αυταχειρισμό που προωθεί η ρωσική προπαγάνδα, φυσικά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση και με την ε, βία, ποια είναι η σύνδεση με τη βία. Και βλέπουμε ότι εξαρτάται από το πώ κινητοποιούν οι δυνάμει αυτέ, οι ομάδε αυτέ τους ε, φορεί του. Η ISIS το κάνει αυτό με τα άτομα που ε, προωθούν το μήνυμα της ε, στην Ευρώπη και προωθούν το γενικότερο μήνυμα και έχουν συγκεκριμένα μηνύματα για τους ακτιβιστές προκειμένου να βγουν στους δρόμους, και να διαμαρτυρηθούν με μη βίαιο τρόπο ή και να επιδείξουν βίαιη αντίδραση. Τύποι λοιπόν ε, κατά των ε, μεταναστών για παράδειγμα που ήρθαν στο μνημείο και στην τελετή των Βρυξελών. Ε, διέκοψαν την τελετή, φόβησαν τον κόσμο και ανάγκασαν τους αστυνομικούς να τους περιορίσουν. Τέτοια λοιπόν φαινόμενα παρατηρούνται και τέτοια προπαγάνδα σπρώχνει τον κόσμο προς συγκεκριμένες ενέργειες. Ε, δεν θέλω να θέσω το ερώτημα του τι είναι χειρότερο, αλλά σε στρατηγικό επίπεδο η ρωσική προπαγάνδα είναι χειρότερη. Θέλουν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ή θελημένα και με ικανοποίηση χρησιμοποιούν τις ροές τις μεταναστευτικές κατά της Ευρώπης προς τον σκοπό αυτό. Υποστηρίζουν το καθεστώς του Ασάντ. Το καθεστώς του Ασάντ είναι η υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη, ε, για το συντριπτική ε, κομμάτι του πληθυσμού που ε, φεύγει από τη χώρα του. Οι Ρώσοι δεν βγαίνουν να λένε όπως οι να βγει ο κόσμος να δολοφονήσει τον κόσμο στους δρόμους. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι η διαφορά μεταξύ στρατηγικής και τακτικής τέτοιας προπαγάνδας. ο κύριος που μίλησε για τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής και της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ Δεν έχει άδικο. Πρόκειται για κοινωνίες ε, που ε, κατεπηγόντως χρειάζονται αλλαγή. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αλλαγή δεν θα συμβεί σε μία νύχτα. Και δεν μπορεί η αλλαγή να προέλθει από τα έξω. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να πείσουμε τις κοινωνίες να αλλάξουν. Και αυτό παίρνει χρόνο και σημαίνει και επένδυση χρόνου και προσπάθειας. Μιλώντας για την προγραφία της βίας. Και οι άλλοι ομιλητές είχαν δίκιο που υπογράμμισαν. Εγώ όσο στον Καναδά είμαστε καταναλωτές των αμερικανικών μέσων, της αμερικανικής προπαγάνδας, που πάντα προβάλλεται ως ο ήρωας και που προβάλλει τους αντίπαλους ως εχθρό με τις χείριστες περιγραφές. Όντως, η προπαγάνδα χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις εποχές, από ομάδες, θρησκευτικέ ομάδες, κατά άλλων θρησκευτικών ομάδων, από πολιτικές ομάδες και το καθεξής. Από οικονομικές ομάδες ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν μίλησα για την προάσπιση των αξιών μας, γιατί πρόκειται για μια μάχη, για έναν αγώνα και σε, στον αγώνα χτυπάνε και οι δύο πλευρές, υπάρχει η επίθεση, η άμυνα. Αυτό γίνεται σε μία μάχη. Ποτέ δεν θα καταπνιχθεί πλήρωση η προπαγάνδα. Είναι αδύνατον αυτό. Η ποινικοποίηση των ιστοσελίδων. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ε, σήμερα στο διαδίκτυο. Δεν είναι δυνατόν πολύ απλά. Θυμάμαι μια συζήτηση στο Ενωμένο Βασίλειο ε, με τον Ήρα μπορούμε να πούμε στους δημοσιογράφους να μην δημοσιεύσουν κάτι. Τότε μπορούσαμε μάλλον. Να περιμένουν δηλαδή για να δημοσιεύσουν κάτι. Τώρα δεν γίνεται πλέον αυτό. Κάθε οργάνωση, κάθε ΜΚΟ, κάθε άτομο ε, περιμένει την επόμενη συντρακτική είδηση. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με τις ιστοσελίδες είναι να τις παρακολουθούμε. Να τις παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε την κίνηση στις ιστοσελίδες αυτές, στις μυστικές υπηρεσίες, το κάνουμε αυτό τσεκάρουμε κάποια άτομα που βλέπουμε ότι εμφανίζονται σε κάποιες ιστοσελίδες, ενώ για παράδειγμα χρησιμοποιούν και μια άλλη διεύθυνση IP όταν μιλάει σε μια άλλη σελίδα. Δεν θα μπορέσει κανείς ποτέ να ελέγξει τις ιστοσελίδες, γιατί θα ανοίξουν την άλλη μέρα από άλλο σερβερ από άλλη χώρα. Το κάνουν και γι' αυτό είναι σε θέση να συντηρηθούν τόσο πολύ για το τελευταίο θέμα, για το θέμα των ημάμιδων που αναφέρατε. Σε ό,τι αφορά τους ριζοσπαστικοποιημένους ημάμιδες, δεν θα ήθελα να θέσω το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει από ένα σημείο και πέρα και ε, ο λόγος προκαλεί μίσος, αντισημετικό, αντιμουσουλμανικό και το μίσος είναι μίσος πάντα για τους ημάμιδες που το κάνουν αυτό. Καμιά φορά απορώ και ενίσταμε. Διαβάζοντα, για παράδειγμα, για τον ριζοσπαστικοποιημένο ημάμι στι Βρυξέλλε που ριζοσπαστικοποιεί και του νέου. Προαγάγει μια ιδεολογία τέτοια στου νέους. Το διαβάζουμε αυτό, διαβάζουμε για τα άτομα αυτά. Διαβάζουμε και για τους νέου που έστειλε στη Συρία. Και μετά θα διαβάσουμε για τους νέους αυτούς που επέστρεψαν από τη Συρία και που έκαναν κάποια επίθεση ή που εμπλέκονται σε κάποιο δίκτυο που οργανώνει επιθέσεις. Άρα έχει νόημα να σταματήσει εξ αρχής αυτή η ριζοσπαστικοποίηση, αυτή η προτροπή προς το μίσος, προς τη βία, προς την μετάβαση στη Συρία και την ε, εκπαίδευση για την ε, εκτέλεση επιθέσεων. Ίσως ε, θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στον επικοδομητικό διάλογο. Θα πρέπει να γίνονται λοιπόν συζητήσεις μεταξύ των ατόμων διαφορετικών ιδεολογιών, αλλά νομίζω ότι ξεπερνάει κάποιος ε, τα όρια του μίσους όταν διδάσκει στα νέα παιδιά να πάνε να σκοτώσουν. Σε αυτό πραγματικά μπορούμε να βάλουμε ένα τέρμα, ένα τέλος. Και η ακαδημαϊκή, ακαδημαϊκή σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, τελείωσε ο χρόνος σας, αν θέλετε να ολοκληρώσετε την πρότασή σας. Ναι, οι ακαδημαϊκοί μπορούν επίσης να τους ε, ε, προκαλέσουν και τα άλλα άτομα και να προκαλέσουν τα επιχειρήματά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε του τρει ομιλητέ μα, Ρέτμα Πομιανόσκης και Σαϊκ. Μίλησαμε για ενημέρωση, μίλησαμε και για προπαγάνδα όπως τονίστηκε, αλλά τώρα θα κλείσει η κυρία Φωτίγιο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ακρόαση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι μια αφορμή να προβληματιστούμε και εγώ να συντάξω την έκθεσή μου. Συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους ότι θα έπρεπε νωρίτερα να τα είχαμε πει όλα αυτά και στην Υποεπιτροπή Άμυνας έχουμε κάνει παρόμοια ακρόαση για το ίδιο θέμα. Ίσως ε, κάπως πιο στενά ήταν αυτά που συζητήσαμε γιατί τώρα φύξαμε ε, δύο πλευρές της ε, στατικής επικοινωνίας. αφενός είδαμε την ρωσική στρατηγική και από την άλλη μεριά συζητήσαμε το ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα ε, που υπάρχει προς νότον από τις χώρες για την ε, ε, ζωσπαστικοποίηση και την στρατηγική που μετέρχονται οι διάφορες Ισλαμικές οργανώσεις είτε μας αρέσει είτε όχι. Και παρόμοια μέσα μετέρχονται και κράτη και μη κρατική φορείς κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Discover this to define and try... Άρα, κάθε κόσμο να δούμε πώς ε, ε, θα βρούμε τα μέσα για να ανασχέσουμε αυτές τις προσπάθειες και θα πρέπει πάντως να ευχαριστήσω την Λετωνική Προεδρία, κατά τη γνώμη μου. Οι συστάσεις της Λετωνικής Προεδρίας ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Θα είναι ένα ορόσημο για να μπορέσουμε να ορίσουμε την αστατική επικοινωνία και να δούμε πώς θα ανασχέσει την προπαγάνδα Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσφατη ανακοίνωσή τη που πήθηνε προς Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Το κείμενο εκείνο μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο μου έδωσε πολλές ιδέες που θα περιλάβω στο κείμενό μου. δύο ενδιαφέρουσε είναι οι παρατηρήσει των συναδέλφων για την αναγκαιότητα του να αξιολογήσουμε και στη συνέχεια να τροποποιήσουμε την οδηγία για τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ σημαντική είναι γιατί ε, τη σήμερα ημέρα υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποια μέσα πάρα πολύ ε, προχωρημένα που σίγουρα θα πρέπει να τα λέμε υπόψη. Πάντως θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτό το οποίο είπε ο τρίτος ομιλητής όσον αφορά το ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους, εκείνους που επιστρέφουν από Συρία, Ιράκ και αλλού. Και ανοιχτά να τους τα πούμε. but, but it may be uh, a real step forward. Αυτό θα είναι ένα ουσιαστικό βήμα πρόοδο. Νομίζω ότι το να καθόμαστε άπρακτοι και να τους παρατηρούμε απλώς τότε χάνουμε την οποιαδήποτε ευκαιρία. Επίσης, συμφωνώ μετά της Αζωφικής Ταξιαρχίας. Βεβαίω και στην Ουκρανία σοβεί διαφθορά. Και ο καθένα βέβαια αυτό το προβάλλει από την τοπική γωνία και τέλος πάντων μετά από με ίσω ίσως δεν είναι τόσο σωστό να κατηγορούμε μόνο μία χώρα που προσπαθεί να ξεπεράσει το δύσκολο σοβιτικό παρελθόν και το κάνει αυτό μόνη της χωρίς βοήθειά μας. Αλλά έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιστραφεί αυτή η πορεία. Ευχαριστούμε κύριε Φωτικαλή Πρόεδρος και σας πενθυμίζω ότι 24 Μαΐου θα στήσουν πρώτη φορά και το θέμα και 26 πέμπτη τροπολογίες και με 100 θα γίνει ψηφορία. Λοιπόν, αναλαμβάνω την Προεδρία. Διότι πρόεδρο και αντιπρόεδροι euh, sont euh, απουσιάζουν. Θα συζητήσουμε τώρα την Τινησία. Έχουμε μελέτη ευρωπαϊκή πολιτική στην Τινησία πριν και μετά την Επανάσταση σαν Επιτροπή. Ζητήσαμε τη μελέτη που συμπληρώνει την έκθεση Καστάλτο. Πριν την παρέμβαση Καστάλτο θα ζητήσω την κυρία Ριμαϊντή, καθηγήτρια διεθνών τραπεζικών συστημάτων στην ανώτατη σχολή, εμπορική σχολή του Μοντρεάλ. Είναι και πρόεδρος της Ευρωμεσογειακής Ενώσεως των Οικονομολόγων και ερευνήτρια ε, στο Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο, επισκέπτρια καθηγήτρια. Είχε την καλοσύνη να αποδεχθεί, να ξανάρθει, να παραστήσει συζήτηση τη έκθεση που θα συζητείτε την ημέρα των επιθέσεων και ξανάρθε σήμερα. Ευχαριστώ κυρία καθηγήτρια που ήρθατε. Να σας δώσω παρεθεί το λόγο και μετά θα καλέσουμε και τον κύριο Καστάλντο να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Τιμή για μένα να είμαι μαζί σας για να μοιραστώ κάποια συμπεράσματα της μελέτης. Θα συνεχίσω την παρουσίασή μου αγγλιστή, διότι η μελέτη έγινε στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ την Επιτροπή σας που με προσεκάλεσε, ούτως ώστε να προβώ σε μια αξιολόγηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Ισία προ και μετά την Επανάσταση. Η Τινησία είναι σε σταυροδρόμι σήμερα. Όχι μόνο πολεμά ενδογενή τρομοκρατία και την εξάγει σε άλλες περιοχές και για μένα που είμαι την ίσια είναι ατυχές για μένα που το λέγω αυτό είναι μια χώρα η οποία ήταν στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την επανάσταση και στην προσπάθεια για δημοκρατία. Σήμερα η νεολαία της είναι απογοητευμένη και παρετείται και πέφτει στα χέρια τρομοκρατικών οργανώσεων. Και κατά την άποψή μου οι τρομοκρατικές οργανώσεις βρήκε πολύ εύθραυστα θύματα. Τα χρησιμοποίησε τα παιδιά αυτά όχι μόνο μέσω προπαγάνδας αλλά μέσω και θρησκευτική χαλιναγώγησης. Μεγάλος κίνδυνος αυτός για μια χώρα όπως είναι η Τινησία που είναι μικρή, πολύ μικρή και μια χώρα η οποία οικονομικά μέχρι την Επανάσταση τα πήγαινε αρκετά καλά. Μετά βλέπουμε σαφώς ότι δεν αρκεί η οικονομία Χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτική, κοινωνική και οικονομική για να ευημερήσει η χώρα και να δώσει στους πολίτες και στην νεολαία ευκαιρίες για απασχόληση και για αξιοπρέπεια. Ως την Ισία αυτή είναι η άποψή μου. Να πάω στη μελέτη τώρα. Τι προσπαθούμε να υπολογίσουμε και να αξιολογήσουμε. Θέλουμε να διαπιστώσουμε Ποια θα είναι η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ενώση και την Ισία στο μέλλον, τι μορφή θα έχει. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτοαξιολόγηση και μέσω διαβουλεύσεων, μέσω εμπλεκόμενων ε, φορέων στην Τινησία, με επαφέ με την κοινωνία των πολιτών, αξιωματούχου τη κυβερνήσεω και σε επαφή με διάφορου φορεί τη χώρα. Η Τινησία είναι πρωταρχικό εταίρο με τι χώρες χώρε από το 1995, όταν υπεγράφει η πρώτη συμφωνία σύνδεση. Μετά κινήθηκε προς τη, ε, προς τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών το 2008 για βιομηχανικά προϊόντα. Είναι η πρώτη χώρα που συνήψε τη συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τεράστια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικής φύσεως. Πολύ σημαντική και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας ήταν αυτή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι βασικός εταίρος της χώρας αυτής. Μετά είχαν προνομιούχο εταιρική σχέση το 2012, η μόνη χώρα, μαζί με άλλες χώρες, όχι από την Νότιο Μεσόγειο όμως. Κρίσιμος εταίρος για μελλοντικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής. Αν δείτε την περιοχή από Συρία μέχρι Λιβύη και μέχρι το Μαρόκο, είναι η μόνη χώρα που ακολουθεί διαδικασία εκδημοκρατισμού και ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση. Δίνει δυνατότητες και δημιουργεί δυνατότητες αλλά και μεγάλα προβλήματα όταν δεν είναι καλά προετοιμασμένη μια χώρα να ακολουθήσει τη διαδικασία που είναι δυναμική. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχουν αβεβαιότητες, σημαντική κίνδυνη προς διαχείριση και προσεκτική εξέταση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως τις είδαμε τα τελευταία τρία χρόνια, υπάρχει συμφωνία για την κινητικότητα. Είναι η μόνη χώρα μαζί με την Ορδανία και το Μαρόκο που γίνεται αυτή η συζήτηση για συνεργασία κινητικής φύσεως για την διακίνηση των ανθρώπων και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου και θέλουμε εμβάθυνση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου που συνήθει το 2015 μαζί με το Μαρόκο συμμετέχει. Και αυτή η συμφωνία υπάρχει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντική για να κατανοήσουμε τι σημαίνει για τη χώρα, για την απασχόληση, τι σημαίνει για τις διαθωτικές προσαρμογές στους διάφορους τομείς που πρέπει να εξετάσει η χώρα. Τα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσω να αναφερθώ στις πολιτικές πριν την Επανάσταση. Πρέπει να καταλάβουμε το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αντιληπτή από τους τινησίους, από την κοινωνία της τινησίας. Νομίζω λοιπόν ότι βάσει της αξιολόγησης που κάναμε περιορίστης ανταλλαγή ε, συμφερόντων οικονομικών ε, πολιτικών συνεργασιών με ένα αυταρχικό καθεστώς που ήταν ε, του προηγούμενου καθεστώτος από την ηγεσία του Προέδρου Μπεν Αλή. Υπήρξε συνεργασία με αυτή την κυβέρνηση που μπορεί να συνοψιστεί με τα εξής πλεονεκτήματα. Ασφάλεια έναντι σιωπής, εμπόριο έναντι ενίσχυσης, ωφέλη έναντι ελευθερίας ήταν τα αντισταθμίσματα έτσι ανέπτυξε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα αυτή πριν από την Επανάσταση. Τώρα όσον αφορά ασφάλεια εν συγκρίση με την σιωπή, η πολιτική συνεργασία σχεδόν αποκλειστικά εστιάστηκε επί της θεμάτων ασφαλείας. Σε κάποιο βαθμό υπήρξε αποσιώπηση των μεταρρυθμίσεων που δεν γινόταν, της προόδου προς τη δημοκρατία. Και καμιά φορά απεκρύπτετο και η επιδείνωση της καταστάσεως. Ήμουν ξανά Είχα έρθει πριν την επανάσταση στο Κοινοβούλιο εδώ, μια-δύο φορέ και θυμάμαι τι είπα. Είπα ότι χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση, οικονομική, πολιτική, κοινωνική. Και αυτό το έλεγα πριν την επανάσταση. Στην πραγματικότητα ήμουν μία από πολλού, ίσω την μειονότητα, τη μειοψηφία επαναφέρθηκε σε αυτό. Είχα πει, α δούμε τα πριν η προσέγγιση ήταν πρώτα τα οικονομικά και τα πολιτικά θα ακολουθήσουν. Όμω οι πολιτικέ εξελίξει ποτέ δεν ακολουθούσαν. Το ξέσπασε η Επανάσταση, το είδαμε. Κατεστράφει η κοινωνική σύμβαση μεταξύ παλαιάς κυβερνήσεω και πολιτών. Τώρα, δεύτερο αντάλλαγμα, εμπόριο εναντί ενίσχυση. Ανοίξτε την αγορά και μετά θα σα δώσουμε οικονομική βοήθεια για να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερο άνοιγμα και φιλελευθερωποίηση χωρίς να εξετάσουμε ρεαλιστικά τις συνέπειες που έχει αυτό στην απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ε, πολλοί, ε, πολλές ε, μειονεκτούσες περιοχές στην Τινησία, ακόμα και στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες υπάρχει αυτό. Κυρίως στην Τινησία εστιαστήκαμε στις Μητροπόλεις και έμειναν πίσω οι άλλες περιοχές. Ήπεθρος, χωριά, ή πόλεις όπως το City που είναι υποανάπτυκτες περιοχές. Η ανεργία των νέων κινείται σε διπλά ψηφία εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι το γνωρίζουν. Τι έγινε? Τίποτα. Μετά, προφανώς, υπήρξε και αμέλεια όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ένταξη. Αμελήθηκαν αυτά. Πολλοί οικονομολόγοι Τη υποφαινομένη συμπεριλαμβανομένη, λέγαμε ότι χρειάζεται μια ισορροπημένη προσέγγιση, ισότιμη, δίκαιη για οικονομική ανάπτυξη. Όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν. Όλοι να ωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια, δεν μιλάμε για 7-8% οικονομική ανάπτυξη στην Ισία. Ήταν ένα απλό 4% επί σειρά ετών πριν την Επανάσταση. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει καλύτερα για τις περιοχές εκείνες που επί σειρά ετών μέχρι σήμερα ε, είναι σε δυσκερή θέση. Τρίτο αντάλλαγμα, ωφέλη έναντι ελευθεριών. Κέρδη έναντι ελευθεριών. Υπήρξε κοινωνικο-οικονομική συνεργασία. Αμελώντας όμως πολιτικές διαστάσεις της κοινωνικής αναπτύξεως. Η κοινωνική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για χώρες ε, που αναπτύσσονται. Κυρίως όταν η πλειοψηφία των νέων και του πληθυσμού είναι αγράμματη. Άρα φιλοδοξία τους είναι να έχουν θέσει απασχόλησης, να χτίσουν τις χώρες τους, αλλά δεν υπάρχει κοινωνική ανάπτυξη σε κάποιες περιοχές και σε κάποιους θύλακες της χώρας. Και ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Η Τινησιακή Επανάσταση έγινε το 2010 Κατεστράφει η κοινωνική σύμβαση με την κυβέρνηση, ξέσπασε η επανάσταση και το κόστος υπήρξε τεράστιο. Υπήρξε επιμόλυνση που επηρέασε και τις άλλες χώρες με παρόμοια προβλήματα. Την νεολαία που είναι δυσαρεστημένη, δεν έχει προσδοκίες και ελπίδες και αυτό ήταν άμεσο αποτέλεσμα της κακής διακυβερνήσεως, κακών κυβερνήσεων, κακών πολιτικών θα έλεγα και ταυτόχρονα κυβερνήσεων και πολιτικών που νομιμοποιούνταν από τη διεθνή κοινότητα. Με την Επανάσταση λοιπόν είδαμε δύο διαδικασίες δυναμικής φύσεως. Δύο διαδικασίες με αβεβαιότητες και κινδύνους και, κάτι, και πολύ σημαντικούς κινδύνους. Εκδημοκρατισμός ξεκίνησε και αποσταθεροποίηση. Δύο παράλληλες διαδικασίες. Μία θετική, ελπίζουμε να κινείται προς σωστή κατεύθυνση, προς εκδημοκρατισμό, προς δημοκρατική χώρα, δημοκρατική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα όμως οι παράγοντες αποσταθεροποίησεως είναι πολύ ισχυροί. Τους είδαμε, τους βλέπουμε. Από τα δεξιά και από τα αριστερά η Λιβύη βρίσκεται σε πόλεμο, η Αλγερία δεν είναι δημοκρατία, πόρα απέχει από κάτι τέτοιο, η Αίγυπτος κάνει άλματα όπου το γυρίζοντας. Και είναι πολύ σημαντικό όπου βλέπουμε συνέχεια να υπάρχουν γύρω ε, περιφερειακές συγκρούσεις και αστάθεια γενική. Πριν την Επανάσταση είχαμε μία μη βιώσιμη σταθερότητα. Όλοι ήξεραν ήταν θέμα ημερών, μηνών ή ετών η καταστροφή της οροπίας. Διονυζόταν ο έλεγχος της κοινωνίας και της οικονομίας. Και βέβαια βλέπουμε ότι υπήρχε υψηλή ανεργία και αυξανόμενες ανισότητες και κοινωνική δυσαρέσκεια. Είχαμε τα αποτελέσματα. Σήμερα τι έχουμε μετά την Επανάσταση. Στα πλαίσια της δικασίας εκδημοκρατισμού και αποσταθεροποίησεως. Ασταθή βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα για τη χώρα είναι ασταθή. Γι' αυτό, γιατί, ποιοι οι παράγοντες σε αυτό. Προφανώς έχουμε τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση πολλών φυλάκων της κοινωνίας, στη διαμόρφωση πολιτικής. Όλοι θέλουν να έχουν λόγο και θα έπρεπε να έχουν λόγο. Προφανώς συμπεριλήφθηκαν τα Ισλαμιστικά κόμματα επί σειρά ετών εξαιρούντο και την ημέρα που τους ήρθε ευκαιρία να αποκτήσουν εξουσία, ξέρουμε τι συνέβη και σήμερα προσπαθούν να διατηρήσουν την εξουσία στο πολιτικό προσκήνιο. Αλλά βλέπω τεράστια προβλήματα να διαφαίνονται, κυρίως διαπιστώνοντας το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, κυρίως στη Λιβύη και άλλες χώρες, όπως το Ιράκ και την αύξηση της ισχύω των τρομοκρατών του Ντάες και άλλων. Υπάρχει τεράστια βεβαιότητα και εξαιρετικές οικονομικές δυσκολίες δυσκολίε που αντιμετωπίζει την Ισία. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο υπέγραψε νέα συμφωνία με την Τινησιακή Κυβέρνηση ύψου 2,5 δι Από πλευρά οικονομική. δεν καταλαβαίνω πώ θα ξεπληρώσει η χώρα τα δάνεια του Νιτάφ. Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να εκδώσει ομόλογα στι διεθνεί αγορέ. Δεν κατάλαβα όμω πώ θα πληρώσουν για τα ομόλογα, για τα κουπόνια αυτό σημαίνει ότι σωρεύει χρέος η χώρα. Ποιος θα πληρώσει με ένα ποσοστό ανεργίας διπλών ψηφίων και η αγορά εργασίας δεν παρέχει ευκαιρίες στους νέους για να εργαστούν. Ποιος θα τα πληρώσει τα χρέη, δεν ξέρω. Τρίτον, τρίτος παράγον για την ασταθή βιωσιμότητα είναι τα προβλήματα λόγω των εντάσσεων στην περιοχή και των συγκρούσεων. Το είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει όλο και πιο πολύ σε ε, πολυτρομοκρατία στην Τινησία, από την νεολαία και από τα χωριά, στα πολύ φτωχά χωριά. Ποιο είναι το μέλλον τους. Ε, ζωφερό. Ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον λοιπόν. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την νεολαία, η προοπτική δηλαδή της ΔΑΕΣ. να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν είναι κάτι αυτό που το διαβάζουμε απλά στις εφημερίδες. Είναι πραγματικό φαινόμενο. Σε ό,τι αφορά την οικονομική πτυχή τώρα. Φυσικά οι εξαγωγές της Τινησίας ε, είναι μεγάλες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά αγαθά. Ε, υπογραφική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Υπάρχει όμως το ε, έλλειμμα σε ό,τι αφορά τους τρέχοντες ισολογισμούς. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την οικονομική κρίση δεν στην Ευρώπη Ασφαλώς οι σχέσεις ε, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση των προϊόντων που εξεγάγει την Ισία, ο βασικό οικονομικό εταίρο είναι οι ευρωπαϊκέ χώρε και κυρίω κάποιε εξ αυτών επλήχθησαν από την κρίση, ιδιαίτερα μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε λοιπόν ε, με σαφήνεια ότι είναι μειούμενη η τάση στις οικονομικές δραστηριότητες της Τινησίας, ιδιαίτερα την περίοδο 2009 2010 αυτό επιδίνωσε παρετέρω την, ε, την ισιακή οικονομία και την ε, έβαλε σε πτωτική πορεία σε ό,τι αφορά τις ε, άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις δεν τις προσελκύει ιδιαίτερο την Ισία και είναι πολύ χαμηλά τα επίπεδα σε σχέση με το ότι προσελκύει για παράδειγμα το Μεξικό από τις ΗΠΑ και από άλλους εταίρους σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και την Ισία, η σχέση τους έχει αλλάξει μετά την Επανάσταση. Υπήρχε σαφέστατα ένα περιθώριο ανάδειξης της σχέσης τους μετά την Επανάσταση. Η διαδικασία εκδημοκρατισμού μπορεί να σημαίνει και σύγκληση με τις ευρωπαϊκές αξίες, ιδιαίτερα αν ε, η πλειονότητα του κόσμου θέλει και έχει φιλοδοξίες για μια σύγχρονη μοντέρνα κοινωνία. Αλλά ούτε αυτό είναι και βέβαιο. Γιατί υπάρχουν και άλλα τμήματα του πληθυσμού που μπορεί να θέλουν πιο πολύ συντηρητισμό, πιο πολύ μουσουλμανικές αξίες. Που κατά τις πρώτες ε, εκλογές Εγώ είδα πόσοι ψήφισαν για Ισλαμικά κόμματα. Κάποιοι μπορεί να τα απογοητεύτηκαν από την κοινωνική και οικονομική απόδοση των Ισλαμικών κομμάτων. Αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει και δεν είναι σαφή οι, οι ισορροπίες. Δεύτερο σημείο, η αποσταθεροποίηση. Η αποσταθεροποίηση λοιπόν συνεπάγεται και ανάγκη υποστήριξη Οι διεθνεί οργανώσει όπω το ΔΝΤ, το Παγκόσμια Τράπεζα και όλοι αυτοί υποστηρίζουν, αλλά υπάρχει και ένα τίμημα και το τίμημα θα πρέπει να το πληρώσουν οι μελλοντικέ γενιέ. Πώ όμω θα το πληρώσουν, είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεθεί επιτάπητος προκειμένου οι θύνοντες ε, στην την νησία. Προτού υπογράψουν ε, για άλλα δάνεια, προτού υπογράψουν άλλες συμφωνίες, να το έχουν υπόψη τους. Οι νέες προκλήσεις για μια διαφορετική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα είναι δύσκολο να επιτευχθεί η συνένεση. Γιατί, γιατί είναι πολλοί οι φορείς που εκφράζουν την πολιτική τους άποψη και είναι μεγάλη η κριτική που ασκείται σε ό,τι αφορά τους τομείς ε, συνεργασίας που θεωρούσαμε ότι είχαν κατηρθεί πλέον μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τενησίας για πολλά χρόνια, όπως για παράδειγμα απελευθέρωση εμπορίου, ασφάλεια, μετανάστευση. Όλα αυτά δεν είναι σίγουρα πλέον σήμερα. Δεν είναι σίγουρο ότι η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερα δυνατή για την Τινησία ιδιαίτερα, αν και η ίδια η Τινήση και οι κυβερνήσει ε, της κοινωνίας των πολιτών διαπιστώνουν ότι προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικά της συμφέροντα. Το συζητάμε αυτό λοιπόν ε, με διάφορους φορείς στην Τενησία ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια ισόρροπη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την πολιτική συνεργασία μετά την ε, Επανάσταση Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε η αντίληψη ότι υποστήριξε πλήρω την δημοκρατική διαδικασία στην Τενησία προσπαθώντας να ενισχύσει τις δημοκρατικές παραδόσεις στην χώρα, αποστέλλοντα ε, αποστολές και τα χρήματα, χρηματοδοτώντας αυτή τη διαδικασία για την, Ισία. Η Ισία λοιπόν τον αναγνώρισε αυτό και την την τον αναγνώρισε αυτό. Και έγινε επίσης μία κίνηση για την ε, περτέρω προώθηση των δημοκρατικών αξιών. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ της ε, ρητορική και της πρακτικής ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές επί τόπου. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη γειτονία, την προώθηση των κοινωνικών συμφερόντων και όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν. Υπάρχει η θεωρία και η ρητορική που είναι καλή και άγια, αλλά η πραγματικότητα διαμορφώνεται διαφορετικά. Θα πρέπει και αυτή να καθιερωθεί και να προσαρμοστεί σε αυτά που χρειάζεται η χώρα σήμερα. Η πρακτική για την ε, ε, πολιτική της γειτονίας εστιάζεται σε θέματα ασφαλείας προς συμφέρον της Ευρώπης και με βάση την ρεσιμότητα. Και για να επανέλθω λοιπόν στο θέμα της ρεσιμότητας, όλοι το γνωρίζετε. Όταν η Τινησία πέρασε στη φάση εκδημοκρατισμού, δεν ε, καταλαβαίνουμε και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή του more for more. Αυτό θα πρέπει να ισχύει ένα χώρα σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία μετά την Επανάσταση. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς μια πιο συνεκτική υποστήριξη σε ό,τι αφορά ε, την χρηματοοικονομική υποστήριξη της Τινησίας. Ε, υπογράμμισε λοιπόν την θέση της ως βασικός οικονομικός εταίρος, να το τονίσουμε αυτό, και υπάρχει και μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμού για την πρόθεση κοινωνικο-οικονομικών εξέλιξεων σε ό,τι αφορά την ε, ανισότητα, σε ό,τι αφορά την ενεργεία. Κινούμαστε λοιπόν προς μια συνεκτική βιώσιμη ανάπτυξη για την νησία. Υπάρχει δηλαδή νέα ανατροπία σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αποκέντρωση, προγράμματα για την αποκέντρωση, προγράμματα για τις μειονεκτούσες περιοχές και το καθεξής. Αλλά όταν διαβουλευόμαστε και με τον κόσμο επιτόπου στην Τινησία, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για την απελευθέρωση του εμπορίου. Ιδιαίτερα σε αυτές τις ευαίσθητες στιγμές της διαδικασίας εκδημοκρατισμού. Ιδιαίτερος για την οικονομία της χώρας. Η εις λοιπόν και συνεκτική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμα επωφελής για τη χώρα, αλλά κοστίζει χρήματα στην ε, παρούσα φάση πρόθεσμα, γιατί υπάρχει ανάγκη προσαρμογή. Άρα σε ποιου τομεί θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσαρμογή και ποιε θα ήταν και οι συνέπειε. για την απασχολησιμότητα σε κάποιου τομεί όπου γίνεται η απελευθέρωση. Τέλο, η κοινωνικονομική συνεργασία μετά την Επανάσταση, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη τη κοινωνία των πολιτών την ενίσχυση των οργανώσεων, των κυβερνητικών οργανώσεων, ε, τι επαφέ με τέτοια άτομα. Και βελτιώνεται η συμμετοχή των οργανώσεων αυτών στον διάλογο για την χάραξη της πολιτικής και στις διαβουλεύσεις. Και υπάρχει πάλι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την διαφυγή εγκεφάλων, το brain drain, σε διάφορου κλάδους. Και θα ήθελα κλείνοντα να πω το εξή. Ποια είναι τα στοιχεία για την βέλτιστη και πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Καταρχά, να βασιστεί η πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνεργασία σε συνεργασίε, σε συμπληρωματικά συμφέροντα, όχι σε αντισταθμίσματα και όχι σε μονομερή συμφέροντα να υπάρχουν μελέτες αντικτύπου και τομεακές και γενικές και διαβούλευση με τους εμπλεκομένους φορείς και θα οργανώνονται διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους φορείς. Ε, επίσης, κατά δεύτερον, διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε την αρχή της ε, ρεσιμότητας και βάση της αρχής ε, της κοινή ιδιοκτησία, της πολιτικής win-win. Τέλος, σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη όλων των ε, φορέων της νησιακής κοινωνίας στη διαδικασία αυτή ε, διαβούλευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και υποθέτω ότι θα δημοσιευθεί γρήγορα αυτή η έκθεση που την έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, λέει ο Πρόεδρος. Και, όπως είπα και προηγουμένως, Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Καστάλτο, που είναι ο εισηγητής μας για τις σχέσεις με την Τινησία στο περιφερειακό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται σήμερα. Ας πάρει το λόγο λοιπόν πρώτος, να μας μιλήσει για την έκθεσή του και στη συνέχεια οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο για να εκφραστούν. Επί της ε, έκθεσης που παρουσιάστηκε, αλλά και επί της έκθεσης του κυρίου Καστάλτο. Φάμπιο Μάσιμο Καστάλτο. Merci beaucoup, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τα χαρά σας βλέπουμε στα νέα καθήκοντά σας σήμερα. Fantastique. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά πρώτον ευχαριστήσω εκ βάθου καρδία την γραμματεία για την εξοχή δουλειά που έκανε και του κοιόδη ηγητές για τη θεσιμότητά του που εκδηλώθηκε από την πρώτη συνάντηση όσον αφορά την εκθεσή μου. Η περίπτωση τη Τινησίας, όπω παρουσιάστηκε, σαφώ από την εμπειρογνώμονά μα είναι θεμελιώδους σημασίας χρήση της μεγίστης προσοχής μας. Και όπως τα είδατε, αναλύοντας το σχέδιο κειμένου, ε, ήθελα να βάλω διάφορες παραγράφους που ε, εμπλουτίστηκαν ε, και θα αλλάξουν μέσω τροπολογιών. 22 Απριλίου είναι η ημερομηνία για τις τροπολογίες. Με τη συνεισφορά σας θα ολοκληρώσουμε το κείμενο. Η δημοκρατική μετάβαση η διαδικασία, η ειρηνική αυτή που έγινε στην Τινησία δεν είναι μόνο ένα θετικό παράδειγμα στον ελληνικό κόσμο, είναι μοναδικό παράδειγμα. Η παγίωση του εκδημοκρατισμού είναι πρωταρχική σημασία και για την ε, σταθερότητα της περιοχής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο ρόλος κοινωνίας των πολιτών και του κουαρτέτου ε, οδήγησαν το 2015 στην απονομή του Βαβίου Νόμπελ. Θέλουμε να ξεπεράσουμε απλώ τη διακήρυξη προθέσεων μέσω τη εκθέσεως. Θέλω να ξεκινήσει μια στρατηγική ώστε την Ισία να γίνει προνομιούχο εταίρους μα για τι σχέσει με το Μαγκρέμπ. Και γι' αυτό σκέφτηκα να διαθώσω το κείμενο χωρίζοντα σε τέσσερα τμήματα. Πολιτικέ και θεσμικέ μεταρρυθμίσει, κοινωνική οικονομική ανάπτυξη, ασφάλεια και άμυνα, κινητικότητα έρευνα, πολιτισμό και παιδεία. Όσον αφορά τι πολιτικέ μεταρρυθμίσει και τους θεσμούς είμαι πεπισμένος ότι είναι θεμελιώδες για μας να υποστηρίξουμε την συνέλευση των εκπροσώπων του λαού που πρέπει να καλύψει την πρόκληση την τεράστια που έχει. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας και της δημοκρατίας, ελήψη πόρων όμως, και να επαναεξεταστεί ισχύουσα νομοθεσία και να ταιριάξει νομοθεσία με τις συνταγματικές αρχές της νέας συνταγματικής χάρτας. Και αυτό ζητούσαμε να υποστηριχτεί η χώρα και η συνέλευση της χώρας. Γράτω της ευκαιρίας για να προθεήσω ε, την ιδέα μιας εβδομάδας για την Τινησία στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήταν ένα σημαντικό δείγμα υποστήριξης και μήνυμα. Ε, θα δίνει ορατότητα στις εργασίες της συνελεύσεως της κυβερνήσεως της Τινησίας και θα δείξουμε πόσο σημασία έχει για μας αυτή η περιοχή και θα χρειάζεται μεταρρύθμιση ο ποινικό κώδικας. Η διαδικασία της αποκεντρώσεως που θα πρέπει να γίνει γρήγορα, αξιοποιώντας τις προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή, χρειάζεται να προωθήσουμε σβέτες πρακτικές για τα ΜΜΕ και να υποστηρίξουμε την πολύ ζωντανή κοινωνία των πολιτών, που ήταν πραγματικός, κινητήρα πραγματικός κινητήρας της Επανάστασης. Και το βασικό θέμα είναι της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως στη χώρα Υπογραμμίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη ενισχύσεων προς την, την Ισία. Πρέπει να ενισχύσουμε το μέσο γειτονίας και χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμός στις προσπάθειες και με τους τοπικούς φορείς. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε αυτή η βοήθεια που θα δώσουμε να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Θεμελιώδες είναι να προσελκυστούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για να δημιουργήσουν απασχόληση. Όπως φαίνεται και από τη μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα, η ανεργία δεν είναι μόνο ένα από τα βασικά προβλήματα, θα έλεγα είναι το βασικό πρόβλημα. Και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και αφορούν την οικονομία, αλλά πρέπει να προωθήσουν και την ανάπτυξη. Και κυρίως θα πρέπει να ευνοήσουν την ένταξη των νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Να επενθυμίσω επ' αυτού και κάποια βασικά σημεία για μας πιο εύκολη πρόσβαση στις μικροπιστώσεις ε, ε, ε, και καταπολέμηση διαφθοράς. Και θα πρέπει μέσω επενδύσεων να μειωθούν τα διάφορα χρέη της Τινησίας που αφορούν διάφορους τομείς της Τινησίας. Χρειάζεται βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να είναι και το κλειδί για την ανάπτυξη της χώρας. Σημαντικό να επενθυμίσουμε τις περιφερειακές ασυμμετρίες που αναφέρθηκαν, προηγουμένως από την έκθεση. Δηλαδή η ακτή, βόρεια και ανατολική ακτή της χώρας έχουν οικονομική ανάπτυξη πολύ πιο μεγάλη από τη νότια περιοχή και η δυτική. Και οι γνώσεις για τη χρήση περιφερειακών πόρων ίσως να βοηθήσουν τη χώρα στα πλαίσια της συνεργασίας με την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Τώρα αφορά την άμυνα και ασφάλεια, βλέπουμε ότι η ασφάλεια έχει αποδυναμωθεί και λόγω της κρισίμου καταστάσεως η οποία επικρατεί στη Λιβύη και οι αλλοδαποί μαχητές, οι τινίσχοι που πηγαίνουν, προσχωρούν στον ΤΑΕΣ μας προβληματίζει. Χρειάζεται και ε, μια αλλαγή μεταρρύθμιση ε, όσον αφορά τις μυστικές υπηρεσίες της ε, περιοχής ε, της χώρας που θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να ισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τη χώρα και με θεσμού τη Ευρωπαϊκή, Ένωση όπως η Ευρωπόλ. Δεν είναι στις τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπόλ θα συνάψει συμφωνίε και συνάπτει συμφωνίες. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, να στείλουμε το Συμβούλιο να εξετάσει το δεχόμενο να υπάρχει δυνατότητα για την Ισία. Όπως υπογραμμίστηκε προηγουμένω από την εισηγήτριά μα, η κοινωνική ένταξη των νέων είναι το καλύτερο μέσο ώστε να παρεμποδίσουμε την στατολόγηση ξένων μαχητών στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Έτσι κόβουμε τις βάσεις στατολόγησης και εμποδίζουμε να εκμεταλλευτούν τη φτώχεια και τον ελληνικό αποκλεισμό αυτές της τρομοκρατικές οργανώσεις και αποφεύγουμε ταυτόχρονα και κάποια επικράτηση κάποια αυταρχικών μέτρων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά την κινητικότητα, υπογραμμίζουμε ότι η συνεργασία υπεγράφει 2014 μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισία είναι ένα πρώτο βήμα προ την κατεύθυνση. Ζητούμε επίση να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των ατόμων από την Τινησία μέσω απελευθερώσεως από τις θεωρήσεις, κυρίως για τους νέους, τους ερευνητές και τους φοιτητές και θα προσέθετα και καλλιτέχνες είναι θεμελιώδη τα προγράμματα τη κυκλική ε, μετανάστευση και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργασία με τα κράτη-μέλη να δράσει δεόντω. Ε, τώρα η συμπράξη, με οι συνεργασίε μεταξύ ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και κοινά προγράμματα και μόνιμη εκμάθηση, εκμάθηση γλωσσών, τεχνολογιών και παιδεία, όλα αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια απάντηση για τον εκδημοκρατισμό τη χώρα, αλλά και για την καταπολέμηση τη ε, ανεργία. Κλείνω με μια έκκληση που απευθύνω πολιτικής χρειάς. Η αξία της βοήθειάς μας προς την Τινησία ξεπερνά κατά πολύ το οικονομικό και δημογραφικό μέγεθος της χώρας. Η Τινησία μπορεί και θα πρέπει να είναι ένα πρότυπο, ένα μοντέλο για όλη την Βόρεια Αφρική και τον Ισλαμικό κόσμο. Σε μια στιγμή όπου η τάση εξάλλου βλέποντας τι γίνεται σε άλλες χώρες είναι αρκετά αρνητική και αντίθετη όσον αφορά αυτή που βλέπαμε εδώ και κάποια χρόνια εν ώψη της ε, Αραβικής Ανοίξεως που βλέπαμε τότε. Αναλαμβάνω, υπάρχει δυνατότητα να διευρύνουμε το οπλοστάσιο οικονομικής υποστηρίξης όπως κάναμε και για την Ουκρανία, να αξιολογήσουμε ε, κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επενδυτικό ταμείο, δηλαδή ε, δεν μπορούμε να έχουμε την εξίσωση την είδα ίσον Κίεβο. Δεν πρέπει να είναι σύνθημα, πρέπει να το αποδείξουμε και πρακτικά. Όχι μόνο για την Ευρώπη, της Μεσογείου, αλλά για όλη την Ευρώπη. Είναι ένα κοινό πρόβλημα, άρα χρειάζεται να έχουμε και κοινή λύση. Στόχος τελικός, απότερο που ελπίζουμε να πετύχουμε σε κάποια χρόνια είναι η δημιουργία μίας προνομιούχας ε, συνεργασίας πολιτικής και όχι μόνο οικονομικής. Το λέγαμε πριν. Κατά παρελθόν είχαμε επικεντρωθεί μόνο επί των τυχών ασφαλεία. Αντιθέτως τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε με μια δημοκρατία που συνάδει με τις αρχές μας και τις αξίες μας τις ευρωπαϊκές. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για να εκμεταλλευτούμε αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Όπως έλεγε και ο Ναπολέον, μπορούμε να κατακτήσουμε έδαφος. Το χρόνο δεν μπορούμε να ανακτήσουμε. Ε, και περνάνε οι μήνες πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτή την ευκαιρία και να το κάνουμε αυτό θα κάνουμε μια ε, για να προχωρήσουμε γρήγορα θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους κύριους συγκητές. Ευχαριστώ κύριε συγκητά. Δεν περίμενα να ακούσω τον Ναπολέοντα στη συζήτηση. Καλό ήταν που τον ακούσαμε. Σας συγχαίρω για την πολύ ισορροπημένη έκθεση που ταιριάζει με τη γραμμή του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή να υποστηρίξουμε τους ίσους φίλους μας σε αυτό το πλαίσιο. Θα επενθυμίσω ότι η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Είναι ένα εργαλείο πολύ καλό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικό ε, σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, πιστεύω ότι καλό θα ήταν να γίνει μια δεύτερη συνάντηση φέτος Αυτή της ε, Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής θα στείλει ένα πολύ σαφές πολιτικό μήνυμα από την πλευρά μας στα πλαίσια της υποστήριξης των νεοχορηγήσεων. Μετά οι πολιτικές ομάδες τώρα θα έχουν το λόγο, οι σκιώδεις εισηγητές. Καταρχάς ο κ. Κέζα που είναι σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. No, Volevo intanto congratularmi, congratularmi con uh, il collega. Θέλω τη φωτογραφία στον Μπροκ. Και συνεργαστήκαμε με τον εισηγητή και τον ευχαριστώ και δημοσία. Ε, εδώ έχουμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις, ε, συγκεκριμένες προτάσεις και πληρότητα. Από πάσης πλευράς προσπάθησε να είναι συγκεκριμένος. Βέβαια, ε, ευχαριστούμε και την ε, καθηγήτρια μας μίλησε για την Τινησία γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό με σοβαρό και συγκεκριμένο τρόπο να ε, επέμβουμε, να λάβουμε υπόψη πόσο έχει η κατάσταση στην Τινησία και άρα θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον εκδημοκρατισμό και να αποφύγουμε την αποσταθεροποίηση. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι σήμερα κάνει βήματα προς την εμπρόση χώρα. Αλλά είχαμε και κάποια δραματικά γεγονότα που έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τη χώρα. Και όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα έχει η χώρα ένα εκατομμύριο Λιβύων. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να εγκαταλείψουμε μόνο τη στη χώρα. Θα πρέπει να πανεύουμε με συγκεκριμένο τρόπο να βοηθήσουμε και αυτό θα είναι προς το συμφέρον όχι μόνο της Τινησίας αλλά και της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει να μην ξεχάσουμε τον, τη γεωγραφική θέση και τη σημασία αυτής για την ευρωμεσογειακή περιοχή. Έχει επομένω σημασία μεγάλη ο δημοκρατισμό και η σταθεροποίηση της χώρας. Και έτσι νομίζω ότι η Ευρώπη θα έχει περισσότερη ασφάλεια. Είναι σημαντικά αυτά που στην έκθεση ο Καστάλου. Συγκεκριμένες κινήσεις. Να κάνουμε και αυτή την νησιακή εβδομάδα. Πολύ ωραία. και πήγαμε και στην ε, χώρα, εξηγήσαμε πως λειτουργεί το δικό μας ε, κοινοβούλιο, οπότε να βοηθήσουμε και την ε, λαϊκή συνέλευση της χώρας να λειτουργήσει. Να βοηθήσουμε και το φθινόπωρο την διοικητική δομή της χώρας και να βοηθήσουμε να εκλεγούν δημοκρατικά θεσμικά οργανά στη χώρα. Και προσωπικά επομένως εγώ θα βοηθήσω και θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην ε, δικαιοσύνη, να γίνουν ε, μεταρρυθμίσεις στην περιφερειακή πολιτική και πρόκειται για ένα έργο το οποίο εμείς μπορούμε να το αναλάβουμε, να βοηθήσουμε με συγκεκριμένα τρόπο να υποστηρίξουμε την, την Ισία. Άρα αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι πολύ σημαντικά για το θέμα πέραν της υποστήριξης για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται βέβαια και οικονομική βοήθεια. Έχουμε αυτά τα 500 εκατομμύρια και ε, μακάρι να μην αργήσει το Κοινοβούλιο και η Ένωση γιατί θα πρέπει στην περιοχή να έχουμε μια σταθερή χώρα, άρα αυτό θα πρέπει να κάνουμε την Τινησία. Είναι θέμα ασφάλειας και άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για με τη Europol. Να μην αδρανίσουμε, να βοηθήσουμε και σε αυτό το μέτωπο τη χώρα. Να βοηθήσουμε την οικονομία της Τινησίας σημαίνει ας ασφάλειας για την Ευρώπη. Αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε ε, κάτι παραπάνω και εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα υποβάλουμε κάποιες ε, τροπολογίες ούτω ώστε να ενισχύσουμε το κείμενο, όχι ότι διαφωνούμε, αλλά για το να ενισχύσουμε πλευρά ε, ασφάλειας. Άρα ήρθε η ώρα τώρα πιο αποφασιστικά να κάνει κάτι η Ευρώπη, κάτι πιο συγκεκριμένο για να υποστηρίξει τη χώρα. Και και εμείς ως ε, Ιταλοί είμαστε δίπλα στη χώρα και ξέρουμε ότι οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Προσοχή να μην χειροτερέψουμε την κατάσταση με το μεταναστευτικό. Και πάλι ευχαριστούμε τον εισηγητή. Αξίζει να κάνουμε αυτή την κίνηση και τον διαπολιτισμικό και διαθεσκευτικό διάλογο. Σεβασμός και για τους χριστιανούς και για τους άλλους. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα είναι θετική αυτή η έκθεση και ελπίζω το Κοινοβούλιο με σοβαρότητα να βοηθήσει τη χώρα ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριος Παντσέρη για τους σοσιαλιστάς. Άλλωστε είναι και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπής για τις σχέσεις μας με τις χώρες Μαγκρέμπη. Σας ευχαριστώ, λέει Μόνο δύο παρατηρήσεις έχω. Πρώτα πρώτα για την έκθεση και κατόπιν τα όσα μας είπε η καθηγήτρια η κυρία Αγιάντη και τη, για τη σχετική μελέτη μας παρουσίασε. Δεν έχω πολλά να πω για την έκθεση και εγώ ευχαριστώ τον συντάκτη, τον Καστάλτο, γιατί όντως Ήταν πολύ επικοδομητική η συνεργασία μας μαζί του. Το κείμενο αυτό είναι μια πολύ καλή αφετηρία, είναι καλά δομημένο και αναλύει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας και αυτό το οποία αναφέρει είναι πολύ σημαντικά. Να, ας πούμε εκεί που λέει τα της ανάκτησης του χρέους, Τη χώρα Να, όλα αυτά είναι βήματα προ τα εμπρό. Και εμεί οι σοσιαλδημοκράτε θα κατεβάσουμε κάποιε τροπολογίε για να τονίσουμε κάποια θέματα που θεωρούμε σημαντικά. Να, Φερρυπίν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς αυτά θα αναδειχθούν στην κοινωνία και επίσης η συμφωνία ελευθέρων εμπορίου θα πρέπει να είναι ασυμμετρικού ή ασύμμετρου τύπου για να ωφελήσει την κοινωνία. Άρα με σοβαρότητα θα πρέπει να πετύχουμε μια σύγκληση όλων των ε, πολιτικών ομάδων στο κοινοβουλίο μας. Τώρα, για την μελέτη θέλω να τονίσω ότι δεν θέλαμε να γίνει απλώς μια συζήτηση εδώ στην Ευρώπη και καταφέραμε το θέμα της χώρας αυτής να αποκτήσει ψηλή προτεραιότητα ακριβώ όπως κάναμε και για την Ουκρανία. Το κάναμε αυτό, δεν πρέπει να το γιατί για μας είναι γιατί πάρα πολύ χρήσιμο. χρήσιμο για τη χώρα, για την περιφέρεια, αλλά και για την Ευρώπη. Έτσι μπορεί ο κόσμος να δει ότι οι προσπάθειες μετασχηματισμού της Αραβικής ε, Άνοιξης ευωδόθηκαν και άρα είναι δυνατόν σε κάποιες χώρες να προωθήσουμε τον εκδημοκρατισμό. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κάποιες θετικές προσπάθειες ανάπτυξης, το οποίο θα ωφελήσει όλες τις πλευρές. Πάντως, να δούμε τι θα γίνει με την έκθεση, να αποφύγουμε πρώτα-πρώτα τον πατερναλισμό. Και επίσης να στερείται κριτικής ε, ε η έκθεση γιατί πάρα πολλές φορές όσον αφορά τον αραβικό κόσμο θεωρούμε, θεωρούν μάλλον ότι είναι δεδομένη η ενίσχυση και η βοήθεια προς τον αραβικό κόσμο Μιλήσαμε για την αρχή more for more. Εγώ νομίζω ότι είναι μια αρχή που θα πρέπει να έχει χρονικό πλαίσιο για την Τινησία. Να μην είναι δαμόκλειο σπάθη, αλλά να είναι κάτι ε, διαρθρωτικού χαρακτήρα και στη δεύτερη φάση να μην έχουμε ερασιμότητα αλλά να έχουμε συνεργασία αμοιβαία πέραν αυτού όταν λέτε ότι πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η βοήθεια, να δούμε και ποια άλλα σημεία. Υπάρχουν επικρίσεις στην Τινησία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Κέζα. Υπάρχει πρόβλημα στην Τινησία σχετικά με αυτό. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε κάποια κίνητρα πολιτικών αποφάσεων και να μην γίνεται ατέρμον συζήτηση χωρίς αποφάσεις. Κάτι άλλο. Η κατάρτιση, η εκπαίδευση των συμπίνων πολιτικών κομμάτων. Να μην στηρίζονται απλώς σε συμφέροντα. Γιατί να κερδίζει ένα κόμμα τις ε, εκλογές και μετά έχουμε τα ε, συμφέροντα που αναδύονται. Θέλουμε κόμματα τα οποία να έχουν κάποια ιδεολογική πλατφόρμα για το μέλλον της χώρας. Οπότε αυτό είναι σημαντικό πρώτα-πρώτα για τη χώρα που έχει παράδοση ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών. Και τελείως ποιος ξέρει πώς θα πού θα πάει η χώρα. Τέλος, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραμελήσουμε γιατί δεν θα πρέπει στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας να έχουμε θενατική ποινή. Γιατί είδαμε ότι δεν θα πρέπει να αναθεωρηθεί η απόφαση της λαϊκής συνέλευσης. Να, τι αιρεσιμότητα θέλω εγώ. Όχι, δεν λέω ότι θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε τα δικά μας στάνταρ στην Τινησία ούτε αλλού. Κανένα δεν θέλει τέτοιε εκλογέ. Αλλά να υπάρξουν κάποιε κόκκινε γραμμέ για μα. Να. πόσο ωφελεί η εν λόγω μελέτη για το θέμα. Δεν ξέρω αν για του συντηρητικού ο κ. Μπασίρη θέλει να πει κάτι. Είναι σκιώδη εισηγητή. Έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κασάλτο για την ε, συνεχτική παρουσίαση της κατάστασης στην Τινησία. Η ε, εκθέση εστιάζεται σε τέσσερα τμήματα ε, και αυτό είναι ευανάγνωστο. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια, ωστόσο, σε ό,τι αφορά τους τομείς όπου έχω την αίσθηση ότι έχουν τη Καταρχάς, για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα της ασφάλειας και της σταθερότητας στην την ισία ανάπτυξη και θέσει εργασία για τον πολίτη. Αυτό θα δημιουργήσει επίσης και ε, δυνατότητες για τους νέους και έτσι δεν θα στρέφονται στην ριζοσπαστικοποίηση. Να τονίσω επίσης των κρατών μελών, τώρα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προώθησης των εμπορικών ε, σχέσεων. Ας ε, ενθαρρύνουμε λοιπόν την ανάπτυξη του, του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να καταπολεμήσουμε την γραφειοκρατία και να προωθήσουμε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η μακροοικονομική αρρωγή λοιπόν με προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και μικροοικονομικά ωφέλη. Δηλαδή, ναι, γέφυρε και αεροδρόμια, αλλά και η εκπαίδευση των ε, δασκάλων, των καθηγητών, η αντιμετώπιση της λεψιδρίας αποτελούν θέματα που αγγίζουν τον τον πολίτη στην καθημερινή του ζωή. Μεταρρυθμίσεις επίσης, για να υπάρχει και συνεκτικότητα στις μεταρρυθμίσεις. Να μην είναι κατακαιρματισμένη η προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων. Να υπάρχει πολιτική δέσμευση του κόσμου επίσης για την ασφάλεια και την άμυνα θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών με την Τινησία για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Αλλά χωρίς σταθερεότητα στη Λιβύη, ας μην το ξεχνάμε, η ασφάλεια στην Τινησία θα είναι κάτι δύσκολο. Η πλαστική επίση μεταρρύθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Σε γενικέ γραμμέ, ο κ. Καστάλτο συμπεριέλαβε τα θέματα που μα απασχολούσαν. Τον ευχαριστώ. Ωστόσο, κάποιε τροπολογίε θα τι καταθέσω για το μίσο που πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί πιο πολύ η προσοχή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Για τους φιλελεύθερους. Δεν είναι ο συζητητή κύριος Λεβάουτμαντς, ο κύριος Κουίτσουκ θα μιλήσει εξ ονόματος λοιπόν των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Ναι. Εξ ονόματο του συναδέλφου, του κύριου, της συναδέλφου κύριου Βάτμαντς, να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Καστάλτο για τι προσπάθειε του και για το γεγονό ότι συναντηθήκε με του κοιότες. Ε, την Ισία είχε μοναδική θέση με την Αραβική Άνοιξη, αλλά είναι τεράστιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ε, ως προς την ασφάλεια. Δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα και να παρακολουθούμε τι γίνεται λόγω της ΔΑΕΣ. Η έκθεση λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Ωστόσο, η Άλτα θα ήθελε να προσθέσει κάποια σχόλια και θα καταθέσει κάποιες σχετικές τροπολογίες. Καταρχά, σχέση μεταξύ τη έκθεσης και της πολιτικής εξέλιξης στο εμπόριο. Θα πρέπει να τονιστεί. Κατά δεύτερον, έχουμε λάβει αξιόπιστες πληροφορίες από πηγές στην Τινησία ότι για την περίοδο 2016-2020 ένας από τους στόχους έχει αναβληθεί μέχρι το τέλη του χρόνου και το Κοινοβούλιο στην Τινησία θα πρέπει να τα εγκρίνει αυτά. Μόλις στα τέλη του μήνα όμως θα γίνει αυτό. και υπολογίσαμε χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς να έχει εγκριθεί η συμφωνία αυτή. Ένα σχέδιο Marshall για την Τινησία. Πιστεύουμε ότι δεν λείπει η χρηματοδότηση από τη διεθνή κοινότητα, αλλά λείπει το όραμα των Τινησιών για το πώς να δαπανίσουν τα χρήματα αυτά. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε την Τινησία προκειμένου να καταφέρει να ξοδέψει τα χρήματα αυτά με το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο για την κοινωνία και τους πολίτες. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Να πούμε δύο λόγια και για την ανάγκη συμφωνίας επανεισδοχής με την, ε, την Ισία. Οι πιέσεις από την συμμετοχή ζωές και παρά το γεγονός ότι έχουμε στρέψει την προσοχή μας ε, σχεδόν αποκλειστικά στην Τουρκία, να κοιτάξουμε και τις χώρες ε, της, του Μαγκρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βερζιά από την και την Με τη σειρά μου και εγώ θα επενέσω τον Φάμπιο Καστάντο, τον συνάδελφο. Έχουμε συνηθίσει να συνεργαζόμαστε. Οι περισσότεροι και με τους περισσότερους σκιώδεις. Ποιος είναι ο στατικικός ρόλος της Τινησίας η σημασία του ρόλου υπογραμμίστηκε από πολλούς. Χρειάζεται ένα σχέδιο Μάρσολ και εταιρική σχέση, πραγματικά προνομιούχα σχέση, πραγματικά ισορροπημένη, που δεν βασίζεται μόνο στα οικονομικά στοιχεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να επιμείνω σε σχέση με αυτά που είπατε και εσείς κυρία καθηγήτρια. Κάποιοι την ίσχυ έχουν σήμερα την εντύπωση ότι η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται περισσότερο προς τα ευρωπαϊκά συμφέροντα από ότι προς τα συμφέροντα της Τινησίας. Αν θέλουμε να αποφύγουμε αν δεν πετύχουμε σωστή ισορροπία, πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι. κάποιες μεταρρυθμίσεις προχωρούν σωστά. Κυρίως διαφθορτικής φύσεως, όπως τις επενδύσεις, η τραπεζική μεταρρύθμιση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του διάφορου τομεί. Είναι σημαντικό να υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ δανείων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δωρεών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αντίθετα από αυτό που είπαν οι φιλελεύθεροι συνάδελφοί μας, δεν πιστεύω ότι οι δωρεές θα πρέπει να δίδονται μετά την Επανάσταση. Δεν δίδονται δωρεές. Το χρέος της Τινησίας αυξήθηκε 20% έκτοτε. Και έπρεπε να δανείζεται από τις σηματοστικές αγορές η Τινησία με επιτόκια πάρα πολύ υψηλά που δεν μπορεί να τα αντέξει η οικονομία της χώρας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν επ' αυτού. Συμφωνούμε τον Φάμπιο και θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να τονίσουμε κάποια σημεία. Δεν διαφωνούμε. Εντάξει, η συλλογή υπογραφών και λοιπά για, τα, τις πρώτες εκθέσεις είναι ένας περιορισμός. Χρειάζεται κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το υπογραμμίσατε και εσείς κυρία μου. Το θέμα των ανισορροπιών μεταξύ περιοχών, μεγάλων μητροπόλεων και άλλων περιοχών πρέπει να καταβληθούν πάνω σε αυτό προσπάθειες και μπορεί να παίξει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσπαθήσει να επανέλθει η ισορροπία διότι και λύσεις των κοινωνικών προβλημάτων μπορεί να βρεθούν μέσω της αποκαταστάσεως αυτής της ανισορροπίας. Μετά ποιος είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν υπογραμμίζεται αρκετά για την ώρα. Σε επισκέψεις έκανε στην Τινησία. Με εξέπλησε η, κοινωνία, η κοινωνική οικονομία τι ρόλο μπορεί να παίξει. Είναι κάτι το οποίο δεν το προωθούμε αρκετά σαν θέμα. Αναφέρθηκα στο χρέος Υποστηρίζω αξιολόγηση του χρέους. Πιστεύω ένα τμήμα αυτού είναι απεκθές χρέος και θα πρέπει να ανακουφιστεί την Ισία από αυτό αν γίνει πραγματικός έλεγχος για το χρέος. Υπάρχουν εκείνες ευθύνες όσον αφορά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Εμείς τοποθετηθήκαμε από αυτού. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την υποστήριξη για τη θέση των πραγμάτων, υποστήριξη του συνάδελφου Παντζέρη όσον αφορά τη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και εκείνο σημείωσε ότι ψηφίστηκε ο νόμος περί τρομοκρατίας και ε, η θανατική ποινή που επιβάλλεται από αυτού, σιωπήσαμε από αυτού, δεν είναι κάτι σωστό. Αρκετοί από εμά θέλαμε να σεβαστούμε την ισορροπία μεταξύ καταπολεμής τρομοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάνω σε αυτό έχουμε μηνύματα να διαβιβάσουμε. Να επιμείνω και επί τριών άλλων σημείων σχετικών. Τεσσάρων. Επιγραμματικά θα τα κάνω αυτά. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα όσον αφορά την αστυνομία, την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Οι ΜΚΟ διαμαρτύρονται συνεχώς για βασανιστήρια με τη διεθνή σημασία που έχει όρος. Το θέμα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό επίσης, κυρίως όσον αφορά προβλήματα που δημιουργούν οι δημοσιογράφοι και blogger, το θέμα της μεταβατικής δικαιοσύνης πρέπει να εξεταστεί. Δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις όπως αυτές που έχουμε με την Τινησία, αν για τα θέματα της μεταναστεύσεως, για τα θέματα μεταναστεύσεως δεν επιμείνουμε, η Τινησία να θεσπίσει κανόνες για τα δικαιώματα των μεταναστών και το θέμα του δικαιώματος ασύλου. Διότι στα εκατομμύρια τόμων που κατέφθασαν από τη Λιβύη υπάρχουν και Λίβοι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε δραματικές συνθήκες. Είναι και το θέμα των ατόμων χωρίς ηθαγένεια, των απάτηδων πρέπει να ρυθμιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε. Υποστηρίζω τις πολιτισμικές ανταλλαγές και αθλητικές. Το θέμα της παιδείας των λαών και της, ε, του συνεταιρίζεστε κλπ. Εγώ μεγαλίδα, είμαι πιο μακριά την Ισία, αλλά έχουμε την Ισία σε εμά. Έχουμε ένα εκατομμύριο την που ζουν στη γαλλική επικράτεια, στο γαλλικό έδαφος και ξέρω ότι αυτές οι ανταλλαγές ε, είναι κάτι ε, πολύ σημαντικό και θα ήθελα να επιμείνουμε από αυτού στην έκθεση και θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίες για να τι λάβετε υπόψη σας αν έχετε την καλοσύνη κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Γιούρεκ ζήτησε και αυτό το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, κύριο Καστάλτρα για τη δουλειά του και για την εξαιρετική εξαιρετικές πληροφορίες που μας έδωσε η κυρία καθηγήτρια. Να πω δύο λόγια. Σύμφωνα με κάποιες ε, πληροφορίες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Open Doors, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια μετά την Επανάσταση υπήρχε ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την ανεξιδοσκία και από τους χριστιανούς, όχι σε νομικό επίπεδο, γιατί δεν εξετάζουμε αυτό, αλλά στην κοινωνική ζωή. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάσουμε το φαινόμενο αυτό και να προσθέσουμε και άλλη μία έκθεση για το θέμα αυτό, γιατί αυτό έχει να κάνει με την ευθύνη των αρμόδιων αρχών που δεν μπορούν να γνωρίσουν το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να ασχοληθούν με την πρόωθηση των αξιών αυτών του σεβασμού κτλ. Γιατί αυτό άπτεται των κοινωνικών σχέσεων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αγγίζει την του χριστιανούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Να καλέσω την κυρία Γιάννη να πάρει το λόγο τώρα. έγιναν κάποια συγκεκριμένα σχόλια του κυρίου Παντσέρη, αλλά αν θα θέλετε να απαντήσετε και στις άλλες παρεμβάσεις, προφανώς έχετε το δικαίωμα να το κάνετε σε τρία-τέσσερα λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας καταρχάς. Νομίζω ότι αυτό που εξαγάγω στο συμπέρασμα από τη συζήτηση είναι πολύ σημαντικό. Η κατάσταση στην Τινησία σήμερα δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να φανταστεί κάποιο. Γιατί καταρχά τα πολιτικά κόμματα αυτά είναι όλα καινούρια. Κάποια έχουν ήδη εξαφανιστεί και κάποια από αυτά δεν κατανοούν ποια είναι η διαφορά μεταξύ πολιτικού κόμματο και οργάνωση κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις ε, ενδεχομένως και να τη χάνουν χειραγώγησης για πολιτικούς ε, στόχους και σκοπιμότητες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το στοιχείο αυτό και πιστεύω ότι ο μοναδικός τρόπος να το πετύχουμε είναι μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της παιδείας. Να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί η διαδικασία και δημοκρατισμό δεν είναι μια διαδικασία που θα πετύχει σε μια μέρα, σε ένα χρόνο, σε μία μικρή χρονική περίοδο. Θα πρέπει να προωθήσουμε την προθυμία των ε, φορέων στην χώρα να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, είναι φυσικά ε, σημείο κλειδί η οικονομική ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, ασφαλώς πολλά άλλα πράγματα επηρεάζονται, αλλά θα πρέπει να δούμε και την ποιότητα της απασχόλησης, το ρυθμό διατήρησης της απασχόλησης και το ρόλο της αγοράς εργασίας για την απορρόφηση της νεολαίας ε, από τα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Αν κοιτάξετε το προφίλ των Αλβαπών μαχητών, η πλειονότητά τους είναι ε, μηχανική τηλεπικοινωνιών, ε, η ε, τεχνολογίες πληροφοριών είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι τελικά αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν να υπηρετούν μια τρομοκρατική οργάνωση, πιστεύοντας ότι αυτή θα τους οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι μακροπρόθεσμη διαδικασία. Δεν παίρνει ένα χρόνο μόνο. Αυτό γίνεται και με το ίντερνετ, με τα κοινωνικά μέσα, και έτσι μπορεί σε πολλές περιπτώσεις ο κόσμος να μάθει αυτά που θέλει. Είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη για τις κυρώσεις. Συμφωνώ. Απόλυτα. Δεν υπάρχει καμία α, υποχώρηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ούτε σε ό,τι αφορά την εφαρμοστική ποινή. Αυτό που αναφέρατε. Και εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να σπρώξουμε τους Ατενίσιους να κάνουν πίσω και να μην ε, υπάρχει σύγχυση με τα θέματα της τρομοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημείο κλειδί αυτό. Υποθέτω ότι οφείλεται σε έλλειψη εμπειρίας. Αυτό το δικαιολογεί. Μια συντηρητική, πολύ συντηρητική προσέγγιση. και για την πρόθεση του φόβου. Σε τελική ανάλυση, αν προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα, νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη γενικότερη κατεύθυνση της απόσυρσης ε, αυτής του μέτρου που καταστρέφει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα της ε, κοινωνικής οικονομίας, της ε, κοινωνία συμπερίληψη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να υπάρχει πολιτική για να προωθηθούν αυτέ οι εξελίξει. Να διδαχθούμε επίση από τι εμπειρίε τη Ευρώπη, όπου η Ευρώπη ήταν πάντα υπέρμαχο τέτοιων εξελίξεων. Όπω σα ε, ξαναείπα, επαναλαμβάνω ότι παίρνουν χρόνο αυτέ οι πρωτοβουλίε. Και υπάρχει πάντα κίνδυνο ε, σε περίπτωση που θα θέλαμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοιε πρωτοβουλίες ε, για την επιχειρηματικότητα και το καθεξή. Δεν είναι απλό. Παίρνει πολύ χρόνο και χρειάζεται πολλά χρήματα. Για όλε τι διαστάσει. μη και το καθεξή. Άκουσα ένα σημαντικό μήνυμα, το οποίο ήταν το εξή. Χωρίς σταθερότητα στην Λιβύη δεν υπάρχει ασφάλεια στην ε, Ισία και συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό γιατί η ασφάλεια και ο μηχανισμό ασφάλεια τη νησίας δεν είναι τόσο ισχυρό όσο θα πίστευε κανεί. Οι Λιβύοι, λοιπόν και οι τριβέ στη Λιβύη προκαλούν μεγάλε αστάθειε. Ιδιαίτερα προ τα νότια τη χώρα. Και αυτό θα πρέπει ασφαλώ να το εξετάσουμε επισταμένω. Μιλήσατε και για το 1 εκατομμύριο εκτοπισμένου από τη Λιβύη που φιλοξενούνται στην ε, Αυτό και πάλι σημαίνει ότι υπάρχει επιπλέον κόστος το οποίο το επιβαρύνει την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και το καθεξής. Η κυβέρνηση το απορροφά. Αλλά για πόσο καιρό και σε τι επίπεδο είναι σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη. Άκουσα και κάτι για σχέδιο Μάρσαλ και δυνατότητα βελτίωσης ή αύξησης της ε, οικονομικής αρρωγής. Ναι, και συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ επιδοτήσεων και δανείων. Αλλά κάτι άλλο που είναι σημαντικό να κοιτάξουμε τον τραπεζικό κλάδο στην Τινησία που βρίσκεται υπό πίεση. Προσπαθούν να εκπαιδεύσουν τις μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν υπάρχει καλά λειτουργούν κλάδο τραπεζικός, είναι δύσκολο να χρηματοδοτούνται οι μικρομεσαίε επιχειρήσει οι μικρέ επιχειρήσει. Φυσικά υπάρχουν οι οργανώσεις μικροπιστώσεων. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και αυτέ έχουν τα προβλήματά του, γιατί βάζουν, για παράδειγμα, υπερβολικά υψηλά επιτόκια. Άρα, καταρχά θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και επισκόπηση των οργανώσεων αυτών και νομίζω ότι η Ευρώπη βάσει των εμπειριών της κατά την οικονομική κρίση μπορεί να βοηθήσει σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των σχεδίων διάσωση και του καθεξής. Ε, θεωρώ ότι την Ισία στην παρουσιαφάση φάση δεν είναι σε θέση να προχωρήσει τις τραπεζικές μεταρρυθμίσεις. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας στη σημερινή συζήτηση. Και τώρα, για να δευτερολογήσει, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Καστάλτο. Ε, ευχαριστώ πρώτα. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι συμφωνώ με το ότι, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική η μεικτή διακοινοβουλευτική επιτροπή και όπως και ο κύριος Παντζέρη και εγώ ε, εργάζομαι σε αυτή την αντιπροσωπεία και άρα θα πρέπει εκεί να δώσουμε προτεραιότητα στην συνεργασία με τη χώρα και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους βουλευτές της χώρας να συνεργαστούμε για συγκεκριμένα θέματα να σας το πω τώρα στα Ιταλικά και οπωσδήποτε να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα ενθερεντικά τους λόγια, για τα επενετικά τους λόγια, για το έργο που επιτέλεσα εις αυτή την πρώτη εκδοχή του κειμένου. Ε, νομίζω ότι είναι ένα που θα μπορέσει μετά να μας δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις διάφορους άξονες του κειμένου και συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που άκουσα για αυτές τις μεγάλες ε, προσπάθειες για την, ε, ε, για την, την Ισία, όπως είπε ο κύριος Σέζα και καλύφθηκε και εκείνο το εκατομμύριο των Λιβύων οπότε θα πρέπει όπως είπα πριν να δούμε το πώς θα ενισχύσουμε την κοινωνική δημοκρατία γιατί ακόμα ή δεν έχει δοθεί ευκαιρία να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του προχωρημένου συνταγματικού συστήματος της χώρας. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στο ευρύτερο τοπίο, όχι μόνο της αραβικής συγκυρίας, αλλά της παγκόσμιας. Επίσης, Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμφωνήσω με τον πρόεδρο Παντζέρη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ σημαντικό θέμα για μας είναι ένας άξονας και εκεί θα πρέπει να ε, στηριχτούμε και να δούμε το πώς θα δώσουμε κίνητρα για την πολιτική ανάπτυξη της χώρας. Θα πρέπει να αναλύσουμε το πώς θα πεμπλακεί η κατάσταση, πώς θα βγει η χώρα από το συνταγματικό αδιέξοδο και πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα δικαιώματα που κηρύχθηκαν με την Επανάσταση που ολοκληρώνει τη διαδρομή της. Σιγά σιγά. Επίσης θα πρέπει να καταδικάσουμε και εμείς εκείνη την ψηφοφορία που όπως αναφέρθηκε θέλει να επαναφέρει την Αττική ποινή και για την τρομοκρατία. Είναι απεχθής η ποινή αυτή γιατί έχουμε τις ε, αξίες μας του, χάρτη ε, των δικαιωμάτων της ε, Οπότε πρόκειται για ε, αυτή τη χώρα η οποία είπαμε ότι θα βγαίνει από την προηγούμενη φάση και θα μπει σε σειρά προτεραιότητας για μας. Επίσης ελαφρώς, δυστυχώς, διαφωνώ ελαφρώς με τον κύριο Κιουτσούκ, δυστυχώς δεν είναι εδώ, ε, μας μίλησε για κάποιους πόρους για την μακροοικονομική ενίσχυση που μας παρουσίασε η ΥΠΑ και εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ίντα. Αφενός είναι αλήθεια ότι θέλουμε να καταβληθούν και πλέον προσπάθειες στη διοίκηση να γίνουν οι σημαντικές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, αλλά την άλλη μεριά η ενίσχυση και οι πόροι που θα ρίξουμε στη χώρα, αν κάτσουμε και ζυγίσουμε τι ε, ε, δανείζεται και τι ε, παρέχεται, όπως είπε η κυρία Βερζιά, θα δούμε ότι πολλές φορές έχουμε τις μεταρρυθμίσεις που προχωρούν όπως λέει και η έκθεση αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι γίνεται, ό,τι περνάει από το χέρι μας γιατί είναι μεγάλη σπουδαιότητα και η, αξία αυτού του προτύπου, αυτού του μοντέλου που θα αναδείξει η ανάπτυξη της ε, Επίσης να προγραμμίσουμε τις ΜΜΕ που είναι πολύ σημαντικές και εμείς ως κίνημα πενταστέρων στην Ιταλία ε, αυτό το αναδεικνύουμε στις διεθνείς μας σχέσεις ε, οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει την κινησιακή οικονομία να μπορέσει να δημιουργήσει απασχόληση και από γεωγραφικής πλευράς Ξέρετε, το, το, το βόρειο άκρο της χώρας είναι πιο πάνω από το νότιο άκρο της Σικελίας, πολύ κοντά στην Ευρώπη. Δηλαδή, ότι πέραν αυτής της γεωγραφικής γειτονίασης, έχουμε εδώ και πολιτισμική, πολιτιστική γειτονίαση. Επομένω, έχει σημασία αυτό το μικρό θαύμα της Επανάστασης και για την περιφέρεια, αλλά και για όλο τον αραβικό κόσμο. Άρα θα πρέπει να πλαισιώσουμε αυτό το θαύμα και την, την ισιακή δημοκρατία να αποφύγουμε πίσω γύρισμα και αντιπανάσταση. Επομένως, εδώ και τώρα θα πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών. θα πρέπει βέβαια να έχουμε τι κόκκινε γραμμέ. Είπαμε για τι μεταρρυθμίσει, για να ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, τώρα θα χαθεί το τρένο το, τρένο, το οποίο είναι ιστορική σημασία. Αυτό το τρένο δεν πρέπει να χαθεί με τίποτα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καστάλτο. Και τώρα τελευταίο που μας ότι έχετε τρεις μέρες για τις τροπολογίε 22 Απριλίου που είναι η πρώτη και κατόπιν θα κάνουμε τη δεύτερη συζήτηση του κειμένου την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου στην Επιτροπή μας και η ψήφιση στην ΑΦΕΔ θα γίνει το 13-14 Ιουνίου και ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Θέλετε κάτι να προσθέσετε όσον αφορά αυτό. Όσον αφορά τα διάφορα, όχι. Κυρίως το πέρα στις ε, συνεδριάσεις και 23 Πέμπτου θα είναι η επόμενη συνεδρίασή μα ή στα 3. Ε, έχουμε όμως και την έκτακτη συνεδρίαση. Έκτακτη, έκτακτη. Ή στο Στρασβούργο. Ή στα 12 Μαΐου. Σημειώστε το.